God morgon och varmt välkomna vill jag hälsa alla till eh, dagen. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Συνεδρίαση αυτή Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φίλων με πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη σήμερα. Για να τη δούμε αυτή την ημερήσια διάταξη. θα κάνω ένα σχόλιο επ' αυτής και θα το σημειώσετε ελπίζω. Μιλάμε για την έκθεση της κυρίας Κράτσα, η οποία συμπεριλήφθη στην ημερήσια διάταξη για να ψηφιστεί. Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες και με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως της κυρίας Κράτσα, θα αναβάλουμε την ψηφοφορία επί της εκθέσεως αυτής. Άρα, σήμερα θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Κράτσα. Θα γίνει λοιπόν συζήτηση και το σημείο αυτό θα είναι το σημείο 7, νέο σημείο 7, μετά τις άλλες ψηφοφορίες. Οπότε σημειώστε το παρακαλώ. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκρισή της. Πάμε στο σημείο 2 ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα σας πω μόνο ότι στο Στρασβούργο στις 9 Μαΐου η Επιτροπή μας θα συνεδριάσει εκτάκτος, οπότε 9 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, συγγνώμη που είναι τόσο αργά η συνεδρίαση που προβλέπετε στο Στρασβούργο, αλλά έχουμε κατεπήγοντα θέματα που πρέπει να ψηφίσουμε. 9 Μαΐου λοιπόν έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής στο Στρασβούργο. Για την τακτική συνεδρίαση στις 25 Μαΐου θέλω επίσης να σημειώσετε ότι θα γίνει συζήτηση τότε με την κυρία Μάργκοτ Βάλστρομ που είναι ειδική σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες και αυτό το οργανώνουμε μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Αυτά από πληροφορίες στα πλαίσια του σημείου 2 ανακοινώσει της Προέδρου. Πάμε στο σημείο 3 για να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων. Η κυρία Κώστα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τη συνεδρίαση με την κυρία Μάλστρομ, αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε με αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τις μετανάστριες γυναίκες και την κατεπίγουσα κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη προφανώς επίσης. Να μιλήσουμε λοιπόν για την κατάσταση των γυναικών σε αυτή τη θέση. Και για τη διάσταση της μετανάστευσης από την οπτική γωνία των γυναικών. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η ευκαιρία, προτείνω, επιτρέψτε μου απλά να το προτείνω. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, πρόταση αυτή, κυρία Κώστα. Διευκρινίζω. Αυτή είναι η Μάργκοτ Βάλστρομ, δεν είναι η κυρία Μάλμστρομ. Η πρώην επίτροπος είναι η κυρία Βάλστρομ. Πάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 31 Ιανουαρίου 2011, 3 Μαρτίου, 24 Μαρτίου 2011. Θα τα βρείτε στο φάκελό σας τα πρακτικά. Αν δεν παραλάβουμε σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Προχωρούμε. Στην ψηφοφορία. Το πρώτο μας θέμα είναι μία έκθεση για την Ειδική Επιτροπή για προκλήσεις του προϋπολογισμού στα δημοσιονομικές προκλήσεις και τη βιώσιμη Ευρώπη για το 2013. Στις 16 Φεβρουαρίου συμφωνήσαμε με τους συντονιστές στη συνεδρίασή μας ότι θα καταθέταμε έκθεση γραπτός επ' αυτού και οι συνάδελφοι κατέθεσαν και πολλές τροπολογίες που τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, η κυρία Γιανακουδάκη. Συγγνώμη, δεν ξέχασα, αλλά έχασα την κάρτα μου. Αυτό είναι χειρότερο. Μια φορά και εγώ μέσα σε δυόμιση χρόνια. Οπότε θα με επιτρέψετε να ψηφίσω διανατάσεως. Κυρία Γιανακουδάκη, μην ανησυχείτε. Κανένα πρόβλημα. Θα σηκώνετε το χέρι και εμείς θα το σημειώνουμε. Εντάξει. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Επένδυση στο μέλλον νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για ανταγωνιστική βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμού. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, για την πέντε. Η έξι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οκτώ υπέρ. Α, όχι, είναι σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα λοιπόν. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτιδό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 15 είναι τα κατά και 10 τα υπέρ. Ούτε κι εγώ έχω κάρτα. Δεν τη βρίσκω τώρα, αλλά θεωρήστε ότι ψήφισα υπέρ. Προχωρούμε. Ψή, τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 καταπίπτει. 11 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεκατρία. Υπέρ κατά αποχές δεκτή έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 14 υπέρ 12 κατά 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ α καταπίπτει η 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 έχει αποσυρθεί οπότε πάμε στην 20 που και αυτή έχει αποσυρθεί 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 14 υπέρ, 12 κατά. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή η τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τελική ψηφοφορία. Άρχεται. πέρασε. Δεκτή 25 εψήφισαν υπέρ και δύο αποχές. Ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία. Το σχέδιο γνωμοδότησης για το μέλλον των κοινωνικών ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Είναι η έκθεση OVIR. Μια πολύ σημαντική έκθεση, καθότι ασχολείται με διάφορες διαστάσεις που ενδιαφέρουν την ε, Επιτροπή μας. Μεταξύ των οποίων η ανάγκη πρόβλεψης μια σειράς μέτρων και πόρων για την μέρημνα των ε, παιδιών. Θα δώσω αμέσω ε, το λόγο στην κυρία Οβίρ για να μας παρουσιάσει τις απόψεις πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Λείπει. Α, εφόσον λείπει ψηφίζουμε. Να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ Κύριε Ταραμπέρα, τι λέτε. Η 12 στο δικό μου κατάλογο πληρο... Ε, έχει αποσυρθεί. Το 12. λάθος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν αποσύρθηκε η 12. Το επιβεβαιώνω αυτό. Μα το ψηφίσαμε το 12 ούτως ή άλλως. 13. Υπέρα. Τροπολογία 13. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 2. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 13 ψήφοι υπέρ 12 κατά. 17 υπέρ. Α, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Για το 17 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 κατά 12 υπέρ. Το σημειώσαμε. Ψηφίζουμε την 20 υπέρ. Διορθώνει. Την 18 ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Για την 18 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτεται. 11 υπέρ, 15 κατά. 21 υπέρ, κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική πρόταση 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 καταπίπτει. Αποσύρθηκε. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 λέει η ομιλήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα πάμε στην 35. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά ας κάνουμε έναν έλεγχο ψηφίζουμε για την 37 τροπολογία 14 14 υπέρ, 13 κατά, άρα εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Παρακαλώ κύριε Οβίρ. Congratulations, Mrs. Ovir. Συγχαρητήρια κύριε Οβίρ, έχει το λόγο. Να πω δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω και κράτησα τις ευχαριστήσεις μου για το τέλος. Όταν ετοίμαζα την έκθεση, ήμουν υποχρεωμένη να ακούω κάποια μηνύματα το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο ήταν πάρα πολύ καλό και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στο αποτέλεσμα αυτό. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Οβίρ. Προχωρούμε τώρα στην δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχή της Ένωσης της περιφερειακής πολιτικής έκθεση επί της ουσίας. Η κυρία Ζαμπόρσκα είναι η υπεύθυνη συντάκτρια γνωμοδότηση. Τη δίνουμε ευθύ αμέσω το λόγο. Εφόσον έχει να κάνει κάποιε παρατηρήσει, έχετε το λόγο, κυρία Ζαμπόρσκα. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην ε, έκθεση αυτή. Κατατέθησαν περίπου 50 τροπολογίες. Ευχαριστώ και για, την, το συμβιβαστικό πνεύμα. Ήταν ένα εκτενέστατο, ευρύτατο θέμα και σε ορισμένες συμβιβαστικές προτάσεις, γι' αυτό είχα βάλει αρνητικό πρόσημο. Καταρχήν δεν ήμουν κατά των προτάσεων αυτών, αλλά οι τροπολογίες θα έκαναν ακόμα πιο εκτενή την έκθεση. Πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες ελήφθησαν υπόψη στο κείμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία και ελπίζω ότι στην Επιτροπή, την αρμόδια επί της ουσίας, η γνωμοδότησή μας θα γίνει δεκτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα.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 Πέρας. Απορρίπτεται. 15 κατά 12 υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 11 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 κατά 12 υπέρ. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. πίπτη 15. Θέλετε όμως να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 14. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 12 κατά και μία αποχή. Οι 15 και 16 καταπίπτουν, επομένως περνάμε στην τροπολογία 17 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, η... καταπίπτει, λέει η πρόεδρος. Όντως καταπίπτει το τρίτο τμήμα της 17. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 26 άρχτη ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται, 28 καταπίπτει, περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. 2. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 1. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκατέσσερις υπέρ, δεκατρεις κατά και μία αποχή. Δύο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ και 4 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Ζαμπόρσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες για σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και να συγχαρώ όλους τους συντάκτες γνωμοδότησης. Ωραία. Προχωρούμε. Το, σημείο, το καινούριο σημείο 7 στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Το σχέδιο έκθεσης για τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Κράτσα. Συγγνώμη, ε, θα ήθελα να σας πω μην θορυβείτε τόσο πολύ τώρα που θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Γυναίκες λοιπόν και διοίκηση των επιχειρήσεων. Τώρα, το υπόβαθρο για την έκθεση αυτή, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι το ύψος, το επίπεδο συμμετοχής στη διοίκηση των επιχειρήσεων από πλευράς γυναικών είναι πολύ χαμηλό και η έκθεση αυτή αποτελεί ουσιαστικά κείμενο μελέτης για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την επιρροή των γυναικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο μετά από την συζήτηση με την Επίτροπο Ρέντινγκ, η οποία συζήτησε το ενδεχόμενο εισαγωγής ποσοστώσεων αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Η συγγήτριά μας έχει το λόγο, η κυρία Κράτσα, και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πίστευα ότι σήμερα θα μπορούσε να ψηφίσουμε ακριβώς επειδή και εσείς είπατε ότι είναι ένα επίκαιρο θέμα το οποίο συζητιέται σε κάποια κράτη τα οποία παίρνουν και πρωτοβουλίες δεν συζητιέται καθόλου σε κάποια άλλα κράτη και επειδή υπάρχει μια πολιτική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πίστευα, επειδή εμείς έχουμε ξεκινήσει πρώτη την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθυμίζω και για σας και για τις αγαπητές συναδέλφους, ότι ήδη από την αρχή αυτής της ε, νομοθετικής περίοδου ε, έθεσα την πρόταση για να κάνουμε αυτή την έκθεση. Σεβόμενοι λοιπόν τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από την Επιτροπή, στην παρουσίαση των τροπολογιών των ε, συμβαστικών τροπολογιών στη συνέχεια πίστευα θα μπορούσε να ψηφίσουμε για να στείλουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα το μήνυμά μας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς την κοινή γνώμη και τα κράτη-μέλη. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν και ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τις συναδέλφους για την καλή υποδοχή που είχε αυτή η έκθεση. είδε από την πρώτη φορά που παρουσίασα τις ιδέες και ανταλλάξαμε τις απόψεις και επίσης για το ενδιαφέρον με το οποίο συμμετείχαν με διάφορες τροπολογίες για να κάνουμε την έκθεση πιο πλήρη ε, και ε, με δυνατό πολιτικό μήνυμα. Προσπάθησα λοιπόν και εγώ στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες να αναδείξω όλες αυτές τις ιδέες. Θέλω να πω ότι οι τροπολογίες που πήρα ήταν πολλές, αλλά εστιαζόντουσαν σε δύο-τρεις παραγράφους, ε, όχι στο σύνολο της έκθεσης και γι' αυτό είναι δύσκολο σε μια συμβιβαστική τροπολογία να μπουν όλες οι λέξεις που περιέχει μια τροπολογία που έχει έλθει από συναδέλφους, αλλά ε, στόχος πάντα είναι να εκφραστεί το μήνυμα παρά οι συγκεκριμένες λέξεις Λοιπόν, προσπάθησα κι εγώ και με την ε, συνεργασία των συναδέλφων που κατέθεσαν τις τροπολογίες να εκφράσω αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες ε, ε, καλύπτουν το πανόραμα της προβληματικής και των μηνυμάτων καταρχάς αναφερόμαστε στις χώρες οι οποίες ήδη έχουν πάρει πρωτοβουλίες ή ήδη έχουν πρωτοβουλίες σε εξέλιξη για να τονίσουμε ότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και πρέπει να ενδυναμωθεί και να διαδοθεί ε, ε, ε, στα, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη μεριά βάζουμε κάποια, θέτουμε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στις προσλήψεις, στις, στην εξέλιξη της καριέρας, στις προαγωγές, συνθήκες που έχουν να κάνουν με την αντικειμενικότητα, με τη διαφάνεια, με την αξιοκρατία, γιατί πιστεύουμε ότι οι συνθήκες αυτές έχουν ηθική βάση, αλλά από την άλλη πλευρά εξυπηρετούν και την ανάδειξη των γυναικών τονίζουμε δε σε άλλη συμβιβαστική τροπολογία την τροπολογία 2 ότι δεν πρέπει ο στόχος ε, του να πετύχουμε κάποια συγκεκριμένα ποσοστά για τις γυναίκες να, να είναι ένα άλοθη για τις εταιρείες να τοποθετούν στα διοικητικά συμβούλια γυναίκες οι οποίες δεν έχουν, ε, ε, κάνει, δεν έχουν απόδειξη της, των ικανοτήτων της ε, καριέρας τόσο στην επιχείρηση όσο και σε έναν άλλο επαγγελματικό χώρο που είναι δεμένος με τις ανάγκες ενός διοικητικού συμβουλίου. Ε, το άλλο που τονίζουμε είναι οι, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν οι επιχειρήσεις με τη δική τους πολιτική προσωπικού, το mentoring, την παρακολούθηση της καριέρας, την ενθάρρυνση κτλ. Ε, σε άλλο σημείο τονίζουμε τη σημασία που έχει η διευκόλυνση της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους άνδρες και τις γυναίκες ε, και μάλιστα έχω εισάγει και την ιδέα ότι αυτό μπορούσε ε, και με την ευθύνη των κρατών μελών να ενθαρρυνθεί με κάποιες με ενισχυτικά έτσι μέσα ε, όπως είναι οι διευκολύνσεις οι φορολογικές. Ε, ε, το άλλο θέμα το οποίο τονίζουμε είναι ότι την ανάγκη του να έχουμε συγκεκριμένα και μετρήσιμους στόχους. Εδώ θέλω να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων όχι μόνο μεταξύ συναδέλφων αλλά και μεταξύ νοοτροπίας κρατών μελών. Ξέρουμε ότι και στις βόρειες χώρες, που είναι χώρες στις οποίες η ισότητα ξεκίνησε να γίνεται πράξη και εκεί υπάρχουν χώρες και μάλιστα με μεγάλο μέρος της κοινή γνώμης που είναι αντίθετο προς, την, προς τα υποχρεωτικά κουότας. Ε, υπάρχουν ε, επίσης ε, άλλες εμπειρίες χωρών που μας λένε ότι προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η έκθεση ανοίγει το δρόμο στην υπευθυνότητα τόσο των κρατών μελών να ενδιαφερθούν για το θέμα και να πάρουν μέτρα όσο και στην υπευθυνότητα των επιχειρήσεων. δεν πρέπει με την έννοια αυτό θέλω να βγει από την έκθεση με την έννοια ότι μπορεί να, μια νομοθεσία να βάλει ένα κουότα ότι οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν των ευθυνών τους. γι' αυτό δίνουμε, ε, ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τα μέτρα που ήδη παίρνουν οι επιχειρήσεις που παίρνουν και ζητούμε και οι επιχειρήσεις να πάρουν μέτρα διότι έτσι δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στις γυναίκες ότι με την υποστήριξη της εργασίας τους ανεβαίνουν και όχι με μια νομοθετική ρύθμιση που θα πάρει η Βουλή, μια, μια Εθνική Βουλή. Ε, προσπαθούμε δηλαδή όλες αυτές οι υπευθυνότητες να φανούν. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έχουμε δύο παραγράφους που λένε για την υποχρεωτική εισαγωγή κουότα ότι πιστεύουμε από τα κράτη-μέλη και να απαλλάξουμε τις επιχειρήσεις από την ευθύνη τους. Λοιπόν, πιστεύω, ε, προσπάθησα να, ε, να είμαι ισορροπημένη και στην ευθύνη φυσικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαφές ήδη έχει αναλάβει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας υπόσχεται μέτρα, αλλά την ευθύνη τόσο των κρατών μελών, επαναλαμβάνω, όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. Και επίσης κάτι άλλο που έχουμε εισάγει είναι ότι επειδή συνήθως αυτά τα μέτρα, τα υποχρεωτικά, όπου εφαρμόζονται και όπου ελπίζουμε να εφαρμοστούν, ε, αναφέρονται σε μεσαίες, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε και μια ειδική παράγραφο για την ανάγκη μιας οδικής, ενός οδικού χάρτη, ενός οδηγού για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν μικρό προσωπικό σήμερα και που ίσως πιστεύουν ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι η ισότητα στα διοικητικά συμβούλια, άρα η ανάγκη επιβίωσης. Και εκεί ε, ζητούμε έναν οδηγό που θα τους δώσει και σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις ε, την θάρρυνση και την ευκαιρία να εισάγουν την ισότητα στις ε, πρακτικές τους. Ε, αυτά είναι έτσι σε γενικές γραμμές τα μηνύματα τα οποία με τη βοήθεια των συναδέλφων έχουν ενταχθεί στις συμβιβαστικές τροπολογίες και ε, ήθελα επίσης να σας πω ότι προσπάθησα να αποφύγω τις επαναλήψεις. Νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος του μηνύματος που θέλουμε να στείλουμε για ένα θέμα που είναι δυνατό στο περιεχόμενο αλλά πολύ περιορισμένο στην έκταση και συγκεκριμένο να κάνουμε μια μεγάλη έκθεση όπου σε κάθε παράγραφο επαναλαμβάνονται τα ίδια θέματα. Ε, μπορούμε να στείλουμε ένα συνεκτικό, να, να φτιάξουμε ένα συνεκτικό κείμενο που περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους, ε, επιστρέψαμε να επαναλάβω, των επιπέδων ευθυνών ε, και της ε, για να στείλουμε ένα μήνυμα συνεκτικό και καθαρό στο, στην κοινή γνώμη η οποία κοινή γνώμη δεν έχει ακόμη αγκαλιάσει με ενδιαφέρον το θέμα αυτό όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί το θέμα των ε, ποσοστώσεων στην πολιτική να το θεωρούν πιο κοντά τους ίσως γιατί κάθε γυναίκα πιστεύει ότι μπορεί σε ένα δημοτικό συμβούλιο της πόλης της σε ένα περιφερειακό συμβούλιο αν όχι στη βουλή αν όχι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να ενταχθεί είναι κάτι απομακρυσμένο από την κοινή γνώμη ανδρών και γυναικών το θέμα των ποσοστώσεων και των υποχρεωτικών μέτρων στα διοικητικά συμβούλια και γι' αυτό πιστεύω ότι η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει αυτές τις παραμέτρους που δείχνει ότι είναι μια υπόθεση και δική μας των ευρωπαϊκών οργάνων των επιχειρήσεων και των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κράτσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αντιπρόεδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα για το πνεύμα με το οποίο αντιμετώπισε το θέμα των γυναικών στα, στην ηγεσία των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να περάσουμε, να κινήσουμε μια κουλτούρα γενικότερα στα 27 ε, κράτη-μέλη. Μια κουλτούρα που δεν δίνει σήμερα θέση στις γυναίκες. Τη θέση που αξίζουν και που αξίζουν απόλυτα δεδομένης της κατάρτισής τους που είναι ακριβώς ίδια με τον ανδρών. Βλέπουμε ότι στο επίπεδο κατάρτισης τα κορίτσια πηγαίνουν τόσο καλά όσο και τα αγόρια. Η επιτυχία αυτή ωστόσο στην εκπαίδευση δεν μεταφράζεται σε επιτυχία στην σταδιοδρομία. Ούτε το βρίσκουμε στο επίπεδο διοίκηση επιχειρήσεων. Καλωσορίζω λοιπόν το γεγονός ότι η κυρία Κράτσα θέλησε στην έκθεση να κουνήσει, να απομακρύνει αυτό το τελείως παράλογο ζήτημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτό το γεγονός σε μια Ευρώπη που διακηρύσει την ισότητα των πολιτών και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μέσω της ε, έκθεσης αυτής θα πρέπει να επιτρέψουμε να αλλάξει αυτή η γενική αντιμετώπιση της θέσης των γυναικών στις επιχειρήσεις, χωρίς φασαρία, χωρίς προξήματα. Τονίζω ένα δεύτερο και υπογραμμίζω ένα δεύτερο σημείο στην έκθεση Κράτσα. Τον βασικό αυτό άξονα για να αλλάξουν οι νοοτροπίες, τον έθεσε ως στόχο χωρίς ωστόσο να χάσει όλα τα μικρά σημεία που πρέπει να αλλάξουν κατόπιν. Νέα διαχείριση σταδιοδρομίας, νέα προσέγγιση της μισθολογικής ισότητας, νέα κινητοποίηση κατά τις φτώχειες, διότι ξέρουμε ότι η οπισθοχώρηση των γυναικών στην επαγγελματική ζωή και στις θέσεις ευθύνης δημιουργούν αποκλήσεις και εξανάγκης φτώχεια μια νέα οργάνωση εσωτερική της δουλειάς. Αν θέλουμε να ανοίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα δεν τελειώνουμε ποτέ. Οπότε έπρεπε να δώσουμε, να βάλουμε ένα στόχο, μια νέα προσέγγιση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε επιχειρήσεις, ώστε οι γυναίκες να είναι πραγματικά ίσες με τους άνδρες. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας κύριε Πρόεδρε θα θεωρεί τιμή της να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει την έκθεση Κράτσα, μια έκθεση που τιμά το Κοινοβούλιο, απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη και εγώ προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε η έκθεση αυτή να εγκριθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις πολιτικές ομάδες, προς ολόκληρο το Κοινοβούλιο, για να μπορούμε κατόπιν να συνομιλήσουμε με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κορνέλησεν έχει το λόγο, παρακαλώ. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της σπουδότητας των ποσοστώσεων. Είχαμε μία συζήτηση για το θέμα αυτό και πολλά από τα επιχειρήματα ακούστηκαν. Απλά θα ήθελα να πω ότι το μόνο που πραγματικά δούλεψε είναι οι συμφωνίες και οι κυρώσεις. Οι θέσει των γυναικών ε, στην ηγεσία ανεβαίνει μισό τα εκατό το χρόνο. μπορεί να περιμένουμε πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να γίνει. Η συγγήτρια είπε ότι το κοινοβούλιο θα έπρεπε να παίξει ηγετικό ρόλο. Ωστόσο, το ρόλο αυτό δυστυχώς τον πήρε, στην πράξη τον πήρε η κυρία Ρέντινγκ. Απείλησε τις επιχειρήσεις και επιτυχώς εκβίασε πιο σωστά τις επιχειρήσεις το να υιοθετήσουν πολιτικές ε, προώθησης των γυναικών στις διοικητικές σχέσεις πριν το Μάρτιο του 12 ή μη. Και δουλειά μας ως κοινοβούλιο είναι να υποστηρίξουμε τουλάχιστον πλήρως τις απειλές της κυρίας Ρέντινγκ, ούτως ώστε να γίνουν ουσιαστικά αξιόπιστες. Η επιχειρηματική κοινότητα ξέρει ότι αν υποβάλει νομοθετική πρόταση θα μπορούσε να τύχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αυτό και θα ήταν πολύ καλό να είχαμε μια έκθεση εξαιρετικά, με εξαιρετικά ευρεία υποστήριξη. Τώρα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ε, των συμβιβαστικών δεν είχα την εντύπωση ότι υπήρχε βούληση συνενετική. Κρίμα. Ε, καλή είναι η αναβολή για να ετοιμάσουμε συμβιβαστικές προτάσεις που θα ικανοποιούν τις ομάδες. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε διατυπώσεις ε, που θα τύχουν ευρύτερη υποστήριξη από την παρούσα διατύπωση. Βεβαίω θα υπάρχουν και κάποια σημεία πολιτική διαφορά και πρέπει να υπάρχουν. Αλλιώ θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Αλλά ας εξασφαλίσουμε ότι στην τέλη ψηφοφορία για την έκθεση θα μπορούμε να ψηφίζουμε επί των διαφορών, εκφράζοντάς τες στην ψηφοφορία. Χαίρο που αναβάλαμε και είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε για να υπάρξει μια εξαιρετική έκθεση υποστηρίζοντας τις απειλές της κυρίας Ρέντινγκ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτριά μας, την κυρία Ρόδη Κράτσα, για την εξαιρετική έκθεση με πολλές προτάσεις, θεωρώ, που βρίσκουν σύμφωνα τα μέλη της Επιτροπής. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στο τέλος της συζήτησης θα υπάρξει ευρία αποδοχή για την έκθεση. Συμφωνώ και με την προηγούμενη ομιλήτρια που είπε ότι πρέπει να δώσουμε ισχυρό πολιτικό μήνυμα και προς την Κομισιόν και να στηρίξουμε σε αυτή τη θεματική την κυρία Ρέντινγκ. Ε, μια πρόταση πολύ χρήσιμη και καλή στην έκθεση είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για τις γυναι... ποσοστώσεις γυναικών, αλλά η κυρία Κράτσα επέλεξε μια πολύ ευρύτερη προσέγγιση ώστε να μπορούν οι γυναίκες να αναπτυχθούν και να έχουν ανέλυξη σταδιοδρομίας. Αυτό απαιτεί πολλές προϋποθέσεις και κριτήρια. Την ευελιξία στον κόσμο της εργασίας που πρέπει να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο. Ιντικές προϋποθέσεις, πλαίσιο, φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων μελών οικογενειών, ε, ένταξη και των ανδρών στην, ε, στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί όλα τα βάρη σε εισαγωγικά να είναι στους ώμους των γυναικών, να τα επομίζονται μόνο εκείνες και οι άνδρες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει πολύ. Στη δική μου την πατρίδα, τη Γερμανία, απέχουμε ακόμα από αυτά. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία σε πολλά σε μας. Πάντως έχω αισιοδοξία ότι θα πιεστεί και η Γερμανία. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σωστή η επιλογή της κυρίας Κράτσα να εντάξει και αυτά τα θέματα, διότι έτσι δημιουργείται ισόρροπη θέση στην έκθεση και αποστέλλεται και σαφές μήνυμα προς την Κομισιόν. Νομίζω ότι θα έχει ευρία αποδοχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κράτσα για την εργασία της και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα. Ξέρω ότι δεν είναι το μόνο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, το ζήτημα των ποσοστώσεων πάντως. Η κυρία Μωράν Σαχτιέ στην Ολομέλεια πρόσφατα έκανε μια πάρα πολύ καλή δήλωση οι ποσοστώσεις είναι ένα αναγκαίο κακό. Πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε τελικά γιατί τα πράγματα δεν κινούνται από μόνα τους. Και μολονότι καταβλήθηκαν κάποιες ε, προσπάθειες και πολλές φορές ε, και οι ίδιες οι ε, ενώσεις εργοδοτών έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες μονομένα στα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε τα ευκραία αποτελέσματα. Και πολλές φορές οι περισσότερες προσπάθειες παραμένουν στο επίπεδο των προσδοκιών. Καθότι λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι, καθότι θέλουμε να αυξήσουμε την εκπροσώπηση των γυναικών, όπου το έχουμε πετύχει αυτό έχει γίνει μέσω δεσμευτικής νομοθεσίας ή μέσω κυρώσεων. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο βλέπουμε ότι υπάρχει η υποχρέωση στη συμμετοχή στις εκλογές, για παράδειγμα, να υπάρχει μια εξορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε επίση στην Ευρώπη, στην Νορβηγία, ότι εκεί πέρα εγκρίθηκε μια νομοθεσία για τις ποσοστώσει, γιατί δεν εκπροσωπόντουσαν σωστά οι γυναίκες στα ανώτατα επίπεδα των επιχειρήσεων. Και ήταν μια δεσμευτική νομοθεσία η οποία δέχτηκε πολλές επικρίσεις, ε, μια νομοθεσία η οποία συζητήθηκε και σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια και βλέπουμε ότι έχουν φτάσει όμως σήμερα στο 42% και ότι υπάρχουν και κάποιε κυρώσει σε σχέση με την νομοθεσία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να εμπνευστούμε από τέτοια παραδείγματα. Η Νορβηγία δεν είναι μια μακρινή χώρα. Και η ίδια η Επίτροπο, η κυρία Ρέντινγκ, είναι υπέρ τη ιδέα αυτή. Πιστεύω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή, να κάνουμε μια συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ταχθούμε υπέρ τη πρόταση αυτή που θα τροποποιήσει τα πράγματα. Είναι το ένα αναγκαίο κακό, σίγουρα δεν ξέρω χρησιμοποιήσετε αυτή τη φράση στι προάλλε Πάντως ε, πιστεύω ότι μόνο μέσω τέτοιων ε, μέτρων τελικά θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, κάποιοι ενδιασμοί, πάντως τα μέτρα αυτά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Κύριε Κώστα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια πολύ. Πρέπει να πω ότι μας έδωσε μια πολύ καλή βάση και έκθεση, επί της οποίας είμαι βέβαιο ότι με τον περισσότερο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ίσως ε, μεταξύ της τελευταίας συνάντησής μας και τώρα είχαμε ως σκιωδών εισηγητών και τώρα δεν είχαμε παρική χρόνο και χρειάζεται ίσως να προχωρήσουμε λίγο πιο διεξοδικά. Πάντως πιστεύω ότι από τις συζητήσεις είμαι βέβαιη μάλλον ότι θα προχωρήσουμε να κάνουμε και ένα ακόμα βήμα μπρο, κοινό βήμα. Να πω δύο πράγματα. Ας πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Καταλαβαίνω, το ξέρω. Και στη χώρα μου ένα τμήμα του γυναικείου πληθυσμού ε, αμφισβητεί, δεν της αρέσει ο όρος ποσοστώσεις και δεν είναι άντρες, γυναίκες είναι. Και για τον εκλογικό νόμο που τέθηκε το ζήτημα υπήρξε αυτή η αντίσταση. Εμείς θέσαμε λοιπόν μεταβατικέ ρυθμίσει και σε αυτό υπήρχε μια κρίσιμη μάζα γυναικών αντίθετη. Να το παρουσιάσουμε λοιπόν με κάποιον άλλο τρόπο και με τις τροπολογίε μας κάπω αυτό προσπάθησε, το είπε και η συγγήτρια. Πρέπει να παρουσιάσουμε το θέμα προς την κοινή γνώμη μεταξύ άλλων, όχι ω ένα εγχείρημα απέτηση συγκεκριμένη ποσόστος, αλλά από μια οπτική άλλη γωνία. Να κάνουμε διάφανη και βάση των προσόντων, διάφανο και βάση των προσόντων, τον οργανισμό τοποθετήσεων, διορισμών, διοικητικά συμβούλια ή οτιδήποτε αλλού είναι. Ξέρουμε ότι τώρα υπάρχει αυτό το All Boys Network. Η νοοτροπία λέει παραδοσιακά πηγαίνουν οι θέσει σε άντρε και αυτό επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει μια εξέταση προσόντων ανδρών γυναικών. Πιστεύω ότι πρέπει να το προτείνουμε υπό την εξή ε, μορφή. Ένα μεγάλο εγχείρημα όπου οι τίτλοι σπουδών, τα προσόντα ανδρών και γυναικών αξιολογούνται, διότι και πολλοί άντρες Πολλοί άντρε αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υποδιάστερη θέση λόγω της αδιαφανούς διαδικασίας επιλογής τους. Εάν προτείνουμε κάτι τέτοιο, με μια μεγάλη προσπάθεια επιβράβευσης των προσόντων και της διαφάνειας, Ξέρετε ότι στους δημόσιους, στους δημόσιους διαγωνισμούς, στους ανοιχτούς διαγωνισμούς, οι γυναίκες δεν χρειάζονται ποσοστό γιατί κερδίζουν. Όπου έχουμε διαγωνισμούς, οι γυναίκες εμφανίζονται σε πλειοψηφία. Όπου υπάρχει διορισμός, εξαφανίζονται. Άρα να ζητήσουμε διαφάνεια, ποιότητα. Αν παρουσιάσουμε το ζήτημα με την, αυτή τη λογική και να λέμε ότι είναι υποχρεωτικό να παρουσιάζεται ανοιχτά το βιογραφικό των υποψηφίων ανδρών και γυναικών, εμέσως ζητάμε ποσοστώσεις. Και αν δεν πετύχει αυτό, πρέπει να, να απαντήσουμε σε μια αντίδραση που υπάρχει και δεν έχει ξεπεραστεί ούτε στη χώρα μου. Δεύτερον, θα ήταν κάπως δηλό από επιτροπής μας ε, εν ώψη και του ανοίγματο που έδειξε η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ να περιοριστούμε σε ένα μικρό βήμα. Πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι ως κοινοβούλιο να απευθυνόμαστε ε, ενώ παρότι στην έκθεσή σου υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα σαφή να τονίσουμε λίγο πιο προωθημένα. Πρώτον, νομοθετική πρωτοβουλία μέχρι το 12 της Επιτροπής που θα μπει σαν ορόσημο. Δεύτερον, να υπάρξει αρχή Δέσμευση των κρατών μελών να εγκρίνουν την αρχή, την αρχή αυτή, αφήνοντα, είχαμε υποβάλει και μια τροπολογία με την κυρία Γκουρμάη, αφήνοντα τα κράτη-μέλη την αξιολόγηση του τρόπου τη δεσμευτικότητα. Αυτή, γνωρίζοντα ότι υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικοί τρόποι παρουσίας και παρουσίαση των επιχειρήσεων. Στην Ιταλία το 85% των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ μικρέ. Άρα πρέπει να βρούμε μέσα και εργαλεία που θα προσανατολίζουν αλλά θα είναι ευέλικτα. Είναι σαφές ωστόσο από την άλλη ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, το χρηματιστήριο εισηγμένες ή όχι, σημαντικές πρέπει να υπάρχει ένας πολύ σαφής δεσμός, μια δέσμευση. Είναι σημαντικό λοιπόν η ιδιωτικες το χρηματιστηριο εισηγμενε η οχι σημαντικες πρεπει να δώσει ένα μήνυμα που θα ενισχύεται από τη δράση του Κοινοβουλίου Κάποιος είπε ότι υπάρχει κάποια... να μην δείξουμε ότι πάμε προς τα πίσω, να δείξουμε ότι υπάρχει και μια συμμαχία και με τα κράτη-μέλη που δουλεύουν αυτό. Και τελειώνω. Εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι η έκθεση Κράτσα δείχνει ότι είναι πιο ανοιχτή σε ένα άλλο ζήτημα, την αύξηση των κάτω προ τα άνω του αριθμού των γυναικών που συχνά δεν προάγονται, ε, δεν αντιμετωπίζουν διακρίσει στη σιδηροδρομία. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν και για τι δύο διαστάσει, όχι μόνο. Πιστεύω ωστόσο ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Οβίρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα που έθεσε το ζήτημα αυτό και που το χειρίστηκε με πολλαπλό και πολυεπίπεδο τρόπο. Έχω μια ανησυχία που αφορά στη δική μου την πατρίδα. στις επιχειρήσεις οι άνδρες και οι γυναίκες τείνουν να εξισούνται, παρόλα αυτά όμως στα συμβούλια των επιχειρήσεων, των εταιριών, επικρατούν οι άνδρες. 2% μόνο είναι γυναίκες στα συμβούλια. Προσπαθούμε πάντα να θέτουμε το θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πολύ δύσκολο. Οι Εσθονοί και άλλοι στην περιοχή τείνουν να πιστεύουν ότι θα αλλάξουν μόνα τους τα πράγματα. Έχουν γίνει αναλύσεις που έδειξαν ότι μισό τα εκατό αλλαγή έχουμε κάθε χρόνο λόγω της αλλαγής νοοτροπίας. Δηλαδή θα χρειαστούν 100 χρόνια μέχρι να έρθουν σε ένα λογαριασμό τα πράγματα. Οι πολιτικοί επίσης αγνοούν ότι το θέμα των ποσοστώσεων ε, δεν ικανοποιεί όλους. Εάν πάμε από πάνω προς τα κάτω θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αντιστάσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπάθησα λοιπόν όταν μίλησα για το θέμα, προσπάθησα να μιλήσω μάλλον για μέτρα παρά για ποσοστώσεις. Το ίδιο εννοώ, αλλά το διατυπώνουμε με υπιότερο τρόπο έτσι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποια μέτρα τα οποία θα κάνουν τα κράτη-μέλη περισσότερο ανοιχτά στο διάλογο, στην αντιπαράθεση. Εδώ οι πολιτικοί και άλλοι στην πολιτική ελίτ μπορούν να συνεισφέρουν πολύ. Τα ΜΜΕ, για παράδειγμα, γιατί θα προβάλλουν το θέμα. Οι γυναίκες σε επιχειρηματικές ηγετικές θέσεις και η αύξηση του αριθμού των γυναικών αυτών αποτελεί μέρος μόνο της όλης διαδικασίας. Εμείς πάντως στηρίζουμε την έκθεση και ελπίζουμε ότι μαζί με την Επίτροπο Ρέντινγκ θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά και δεν θα χρειαστούν έτσι 100 χρόνια για να γίνουν περισσότερο ορατές τις επιχειρήσεις οι γυναίκες. Επίσης, μια άλλη στατικιστική μοναδική σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι ότι το 2009 το 70% των πτυχιούχων των πανεπιστημίων στην Εστονία ήταν γυναίκες. αυτοί από τους διδακτορικούς φοιτητέ πάνω από το 60% είναι γυναίκες. Όμως σε ηγετικέ θέσεις εξακολουθούμε να έχουμε ένα 20-30% γυναίκες. Διάβασα ε, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθε από μια ευφυή e e γυναίκα η οποία είπε ότι δίκτυα. Ε, που είπε ότι ε, περισσότερο ε, αρέσκονται οι, ε, να έχουν άνδρες σε ηγετικές θέσεις όπως ε, και σε κόκκινες, ε, ε, οι άνδρες αρέσκονται και στα κόκκινα σόρουχα. Já bych chtěla eh, konstatovat, eh, že eh, už původní návrh zpravodajky. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μας άρεσαν οι προτάσεις της εισηγήτριας. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του Σκιώδους ε, από την ομάδα ECR. Συμμετείχα και στην αρχική συζήτηση και η αρχική πρόταση μου φάνηκε πολύ ισορροπημένη, αν και ορισμένες από τις τροπολογίες μας δεν υιοθετήθηκαν 100%. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες εκθέσεις, δεν είναι πρόβλημα. Γι' αυτό θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε σήμερα την έκθεση. Τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες τις έχουμε μελετήσει και υποθέτω ότι όπως και άλλοι ομιλητές διαπίστωσαν πολιτικές ομάδες και οι ιδέες τους αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πολιτικές στάσεις. Ίσως αυτό δυσκολεύει την επεξεργασία μιας ε, συμβιβαστικής λύσης. Πάντως πιστεύω ότι παρόλα αυτά η συγγήτρια τα κατάφερε ιδιαίτερα καλά και γι' αυτό θα είμαστε έτοιμοι σήμερα να ψηφίσουμε την έκθεση. Αφού κάναμε κι άλλη συζήτηση. Θα ήθελα κι εγώ στα πλαίσια αυτά να τονίσω ότι εξακολουθώ να είμαι πεπισμένη ότι στην έκθεση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να γίνουν δεκτές από τα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι από την Τσεχία. Η τσεχική δημοκρατία, εις ό,τι αφορά την εκπροσώπηση σε δημόσια αξιώματα και σε ηθήνουσες θέσεις, η Τσεχία δεν βρίσκεται και στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής ε, ε, κλίμακας. Όμως, αν γίνει η δημοσκόπηση, τότε οι γυναίκες στην Τσεχία λένε, οι ίδιες λένε ότι είναι κατά της εισαγωγής ποσοστώσεων και ότι το πιο σημαντικό για εκείνες είναι το πώς θα δώσουν μάχη για να κατακτήσουν με το σπαθί τους τη θέση τους. Με άλλα λόγια, πώς θα λύσουν τα προβλήματα του νοικοκυριού, της φύλαξης των παιδιών και πώς θα τα συμβιβάσουν αυτά με τη δουλειά τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο βαθμό που δεν υπάρχουν αρκετά κέντρα φύλαξης των παιδιών που να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους εκεί οι γυναίκες και να θεωρήσουν ότι είναι καλή η φύλαξη, το επίπεδο δηλαδή. Θα μπορούσαν αυτά τα κέντρα φύλαξης να οργανώνονται από την επιχείρηση, από το, το Δήμο, του ή από το κράτος. Ε, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλιώς τι σου κάνουν οι ποσοστώσεις. Δεν θα πείσουν τις γυναίκες να πάνε στην ε, επιχείρηση και στις διοικητικές θέσεις ε, εφόσον δεν έχουν λύσει τα άλλα προβλήματα. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα και ξέρουμε τι σημαίνει να συμμετέχει κανείς σε νυχτερινές ε, συνεδριάσεις. Εγώ ξέρω από τη δική μου εμπειρία τι συμβαίνει σε τέτοιου είδους ε, ε θέσεις. Άρα λοιπόν η συζήτηση για τις προσωστώσεις δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ. Μάλλον πρέπει να μιλήσουμε για ένα πλέγμα μέτρων που χρειάζονται ούτω ώστε να βοηθηθούν οι γυναίκες να προχωρήσουν σε μια ανέλυξη της, σταδιοδρομία του της σταδιοδρομίας τους εφόσον το θέλουν. Τέλος, σα είπα, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτή την ισορροπημένη έκθεση όπως θεωρούμε, αλλά θα εξακολουθήσουμε και να συνεργαζόμεθα και να δούμε ποια ε, πορεία θα ακολουθήσει η έκθεση αυτή. Θέλω να ευχηθώ στην εισηγήτρια να ε, φάσουμε σε ένα θετικό και καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τη σκληρή δουλειά της ε, Ρόδης. Επιτρέψτε μου μια σύντομη παρατήρηση. Το χειρότερο μήνυμα θα ήταν η έκθεση αυτή και η όλη ιδέα να αποτύχουν επειδή για ένα κόμμα ε, τα μέτρα που προτείνονται είναι λίγα και για κάποιο άλλο είναι υπερβολικά. Έτσι λοιπόν σας ζητώ να ξανασκεφτείτε τις πιθανές συμβιβαστικές λύσεις ώστε να αποστείλουμε αξιόπιστο και βαθύ και τεκμηριωμένο μήνυμα. Γιατί μέσα από μια μάχη για τις λέξεις μπορεί να χάσουμε σε ουσία. Έχω την εντύπωση ότι οι συμβιβαστικές λύσεις γύρω από στόχους και ποσοστώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Ακούσαμε ότι δεν ισχύουν τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη μας. Επίση υπάρχουν διαφορές μεταξύ ομάδων της κοινωνίας. Ακόμα και μεταξύ γυναικών οι ποσοστώσεις δεν γίνονται 100% αποδεκτές. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε μια άλλη διατύπωση η οποία θα μπορέσει να σπρώξει προς τα μπρος την όλη ιδέα. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις κατάλληλες για την προβολή του μηνύματος. Διότι αν αποτύχουμε στο μήνυμα που θα στείλουμε θα ανασταλεί ολόκληρη η προσπάθειά μας. Και όχι μόνο η δικά μας, αλλά και η προσπάθεια της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ζωμέβα έχει το λόγο. Τέσσερις βασικές παρατηρήσεις. Πρώτον, για το πλαίσιο. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία. Είναι προφανές, διότι οι χειρονομίες και οι λέξεις Επιτρόπου μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαφορετική από ότι αν ε, ήταν διαφορετική η θέση της Επιτρόπου. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή και να βάλουμε το Κοινοβούλιο πρωτοπόρο, όχι πίσω στη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Δεύτερον, ποσοστώσεις. Το θέμα των ποσοστώσεων, με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι ίσονος σημασίας. Είναι ένα αναγκαίο μέτρο, αλλά ανεπαρκές. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι το θέμα του, της τοποθέτησής της. Αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη. Ταυτόχρονα είναι απόλυτα ανεπαρκές μέτρο και αυτό πρέπει να το παρουσιάσουμε. Τρίτον, για να μπορεί η συζήτηση αυτή να έχει νόημα συνολικά, να μην επικεντρώνουμε δηλαδή την προσοχή μας μόνο στο θέμα των ποσοστώσεων, είναι αναγκαίο να εξετάσουμε πώς και με ποιο τρόπο θα αποτιμήσουμε την επαγγελματική δραστηριότητα. Και το πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχουν κλάδοι επαγγελματικοί που θεωρούνται κατώτεροι, κλάδοι που καλύπτονται περισσότερο από γυναίκες και επαγγελματικοί κλάδοι που θεωρούνται πολύ καλοί, με πολλά προσόντα ή που θεωρούνται ότι έχουν πολλά προσόντα και που είναι αυτοί οι κλάδοι που κατά βάση καλύπτουν άνδρες. Η πρόκληση είναι να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Γιατί είναι πιο ποιοτική η δουλειά του διευθυντή ή του επιχειρηματία ή του χρηματιστή από το έργο που κάνει ε, μια, κάποιος στη δραστηριότητα μέρημνας. Γιατί να μην πούμε ότι και οι δύο τομεί είναι θεμελιώδεις ε, δραστηριότητε, Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε στην διαμόρφωση της εκπαίδευση, της ε, κατάρτιση, ούτω ώστε να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών σε παραδοσιακά ανδρικούς χώρου, αλλά και ταυτόχρονα μεγαλύτερη παρουσία των ανδρών σε χώρου παραδοσιακά γυναικείους. Στη συζήτηση λοιπόν η ποσόστοση θα πρέπει να είναι τμήμα μιας ευρύτερης ε, περισυλλογής, ενός ευρύτερου προβληματισμού που να μην λέει μόνο γυναίκες στις επιχειρήσεις αλλά και περισσότεροι άνδρες σε άλλους χώρους για τους οποίους θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν προσόντα. Τελευταίο ζήτημα. Το θέμα δεν είναι θέμα επιχειρήσεων που πρέπει να λύσουν οι επιχειρήσεις αλλά που πρέπει να το δούμε κοινωνικά. Και γι' αυτό ως κοινωνία πρέπει να διαμορφώσουμε τους μηχανισμούς, ούτω ώστε οι επιχειρήσεις ως ένας επιπλέον παράγοντας στο παιχνίδι αυτό να μπορέσουν να αναλάβουν δράση. Παράδειγμα, για να σας δω το πώς, τη συζήτηση για την άδεια πατρότητας. Ενώ είναι πιο προβληματικό για μια επιχείρηση να προσλαμβάνει γυναίκα, διότι μπορεί να μείνει έγκυος και άρα να είναι στο κρεβάτι μήνες και... από ότι έναν άντρα που δεν θα είναι έγκυος, δεν θέλω ότι να έχει το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα, που δεν θα είναι έγκυος, θα είναι πρόβλημα η επιλογή για την επιχείρηση. Εάν εμεί θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι ευθύνη των γυναικών, αλλά και οι άντρες, οι πατέρες η συγκεκριμένη περίπτωση έχουν ευθύνε. και άρα οι επιχειρήσει θα γνωρίζουν ότι τη στιγμή τη πρόσληψης πατέρα ή μητέρα και στι δύο περιπτώσει, θα χρειαστεί το ζευγάρι αυτό να αντιμετωπίσει μία απουσία, εξαφανίζεται το πρόβλημα. Πώς με νομοθετικά μέτρα να λέμε ότι η άδεια πατρότητας δεν είναι θελούσιο περιορισμένο δικαίωμα, αλλά ως κοινωνικό μέτρο, με νομοθετικά λοιπόν υποχρεωτικά μέτρα, αλλά και με δημόσιους πόρους. Απαιτεί επενδύσεις του δημοσίου σε συστήματα μέρημνας που θα επιτρέπουν σε άντρες και γυναίκες να συμφιλώνουν τις δύο διαστάσεις. Τελευταίο ζήτημα. Ωράρια. Χρόνος. Η, η ορθολογική χρήση του χρόνου είναι μια συζήτηση ευρωπαϊκού επίπεδου. Άλλο χρόνο στη Μεσόγειο, άλλο στο, στη Σκανδιναβία. Το θέμα του φωτός. Αλλά το να εξορθολογήσουμε τις ώρες εργασίας ούτω ώστε να μην ξεκινούν όλοι την ίδια ώρα και να τελειώνουν την ίδια ώρα. Να συνδιαλέξουμε τον χρόνο δουλειά με τον χρόνο αναψυχία. Να κλιμακώσουμε τι επαγγελματικέ δραστηριότητε, επιτρέψει σε περισσότερε γυναίκε να μπορούν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων και περισσότερου άνδρες να ασχολούνται με άλλα ζητήματα που δεν είναι διευθυντικά. Όλα αυτά τα ζητήματα, αν τα δούμε και ήδη εμφανίζονται στι ιδέε αυτέ κάπου στι εκθέσει μπορούμε να δούμε το ζήτημα των ποσοστώσεων από μια πολύ πιο σφαιρική προσέγγιση και να μην μιλάμε μόνο για το αν θα πρέπει να έχουμε 2, 3, 4, 5 γυναίκες σε, σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Αν την κάνουμε τη συζήτηση σε, σε σφαιρικό επίπεδο, θα δούμε ότι κλάδοι σε χώρες όπου πιο δύσκολες, ε, είναι πιο δύσκολο, υπάρχουν περισσότερες επιφυλάξεις, να καταλάβουν τη συζήτηση. Βεβαίως, οι συνθήκες είναι αυτές που είναι. Πρέπει να εκπαιδευτούμε το ότι η κυρία Ρέντινγκ έχει μια στάση παρόμοια με αυτή που εμείς οι περισσότεροι θέλουμε, πρέπει να μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε ως εμπροστοφυλακή, όχι ως οπισθοφυλακή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο, η Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συμφωνήσω κι εγώ με τις ευχαριστίες όλων των συμφωναδέλφων ε, προς την, για το θέμα της έκθεσης αυτή. Πραγματικά στο ζήτημα αυτό είμαστε όλοι δίπλα, όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε μαζί για έναν κοινό στόχο. Χωρίς πολιτικές ε, διαφορές, ε, το έλεγε και η κυρία Μπάουερ προηγουμένως, το σημαντικό είναι να περάσουμε το μήνυμα το Κοινοβούλιο, η Ένωση πρέπει να περάσει ένα μήνυμα για τη σπουδαιότητα των ποσοστώσεων που έχουν σήμερα και που θα έχουν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο και έχουν δημόσια παρουσία, δημόσια ιδιοκτησία, αλλά και στην πολιτική. Εγώ ε, μιλώ ως Ιταλίδα. 10% των δημάρχων στην Ιταλία είναι γυναίκες, ένα στις, μία στις δέκα. Άρα χρειαζόμαστε γυναίκες στα δημοτικά συμβούλια. Επανερχόμενοι λοιπόν στα λόγια της κυρίας Μπάουερ, ε, από αυτό προκύπτει η σπουδαιότητα του μηνύματος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ένα θετικό μήνυμα, ιδίως υπό το φως των δυσκολιών των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική προς ορισμένα κράτη-μέλη που δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες, δε, μεγάλες που δείχνουν την τροτότητα των ευρωπαϊκών συνόρων κάποιων κρατών μελών. Θετικά μηνύματα λοιπόν. Θετικά μηνύματα που περνούν μέσω της ενεργοποίησης μέτρων εφαρμόσιμων και πρακτικών και ελπίζω οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν την τροπολογία μου για ειδικέ φορολογικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις εκείνε που επιτρέπουν σε γυναίκε να συνδιαλέξουν χρόνο οικογένειας, χρόνο δουλειάς. Όλες λοιπόν υποστηρίζουμε την έκθεση Κράτσα που πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά επίκαιρη και εξαιρετικά αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Καλημέρα και ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχά την κυρία Κράτσε για την έκθεσή της. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό και θεωρώ να πω πολλά πράγματα. Πρώτον, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πρωτοπόρο πρέπει να έχει ηγετική θέση. Δεν θα ήταν σωστό πολιτικά και κοινωνικά να υπάρξουν κράτη που θα ξεπεράσουν τι πρωτοβουλίε που θα μπορούμε να εγκρίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν χώρε, η Νορβηγία, εγώ είμαι Ισπανίδα και προέρχομαι από μία αυτονόμη περιφέρεια που το 2005 υιοθέτησε ένα νόμο με ισορροπημένη, για ισορροπημένη παρουσία γυναικών και στους εκλογικούς συνδυασμούς και στα διοικητικά συμβούλια. Δεύτερον, Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε την πρωτοπορία, διότι πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε. Και το θέμα είναι ευαισθητοποίηση των κρατών. Πριν εγκριθεί ο νόμος που ανέφερα το 2005, εμείς κάναμε μια έρευνα μεταξύ του πληθυσμού για να δούμε αν ε, θεωρούσε ότι οι γυναίκες έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα, είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. Και μετά από πολλά χρόνια δουλειά, η κοινωνία με ποσοστά που έφτανε σχεδόν το 80% ήταν υπέρ τη έγκριση των ποσοστώσεων και στην πολιτική και στα διοικητικά συμβούλια και να θεσπίζει ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για άντρες και γυναίκε. Έχουμε λοιπόν ρόλο ηγετικό και ρόλο ευαισθητοποίηση. Μετά, να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Ρομέβα την άποψη ότι το θέμα δεν είναι απομονωμένο. Δεν μπορούμε να συζητούμε μόνο για την αντιπροσώπευση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, χωρί να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση γιατί τι γίνεται με τι άδειε μητρότητα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούμε ακόμα κατά πόσον ένα άτομο που παίρνει άδεια πατρότητας ή μητρότητας θα λάβει μισθό ή όχι για την περίοδο αυτή. Δεν έχει λογική και δεν είναι συνεκτικό με τα μέτρα που πρέπει να εγκρίνουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συνέπεια σε όλες τις πρωτοβουλίες που μας απασχολούν. στόσεις. Πριν 20 χρόνια εγώ δεν ήμουν υπέρ των ποσοστώσεων και έμαθα ότι όσες περισσότερες ευθύνες παίρνουν οι γυναίκες τόσο μεγαλύτερη ανισότητα αντιμετωπίζουν. Άρα πιστεύω τώρα ότι είναι αναγκαίο οι ποσοστώσεις και συνέβαλαν τουλάχιστον στη χώρα μου και στην περιφέρεια από όπου προέρχομαι στην βελτίωση της θέσης των γυναικών. Να έχουν δηλαδή 53% στο βασικό κοινοβούλιο παρουσία οι γυναίκες. Τίποτα άλλο, αλλιώ δεν μπορούσε να είχε επιτευχθεί. Η κοινωνία το βλέπει σήμερα σαν κάτι απόλυτα φυσικό. Έξι χρόνια μετά την έγκριση του νόμου που σας είπα. Επιπλέον πρέπει να μπορούμε να περάσουμε και ένα θετικό μήνυμα. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις που λένε ότι οι πιο καινοτόμες και ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρήσεις σήμερα είναι εκείνες που συμπεριέλαβαν μια ισορροπημένη παρουσία γυναικών στους χώρους ευθύνης τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ικανοί να πουλήσουμε αυτό το θετικό μήνυμα. Πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε ειδική προσπάθεια από τα μέσα επικοινωνίας για να προσπαθήσουν να πουλήσουν θετικές εικόνες, θετικά νέα. Μία αυτοκριτική τώρα οι επιχειρήσεις μας παρατηρούν. Και τι βλέπουν στο Κοινοβούλιο και στην ευρωπαϊκή πολιτική, ότι άντρες είναι επικεφαλής. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ποιος είναι ο μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ποιοι είναι οι ηγέτες των κοινοβουλευτικών ομάδων στο σώμα. Πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική λοιπόν. Είναι λογικό λοιπόν, μας βλέπουν οι επιχειρήσεις. Τι θα τους πούμε, κάντε αυτό. Θα μας πούν, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που ζητάτε από μας; Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να την αντιμετωπίσουμε αυτή την, αυτοκριτική. Την αυτοκριτική. Δείτε, προεδρίες επιτροπών. Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι το κοινοβούλιο αυτό, και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, το κοινοβούλιο αυτό επαναλαμβάνει και αναπαράγει τα κοινωνικά στερεότυπα. Οι γυναίκε ασχολούνται, να δείτε εδώ, σήμερα, με λίγε τιμητικέ εξαιρέσει ανδρών. Ποιο ασχολείται στις πολιτικές ισότητε. Σε μια άλλη επιτροπή βιομηχανίας μεταφορών βλέπετε ότι η αντιπροσώπευση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Να απαντήσω τώρα και στον κύριο Ρωμέβα που έλεγε να επενδύσουμε στην επαγγελματική αξία. Οι γυναίκες δεν μάθαμε κάτι που το κάνουν πολύ καλά οι άντρες. Μια γυναίκα που μαγειρεύει όλη της τη ζωή είναι μάγειρας. Όταν ένας μάγειρας είναι καλός γίνεται σεφ και λέμε να ηγέτες, γαστρονομική, ηγέτες. Πάλι άντρες. Και αυτό γίνεται παντού. μια γυναίκα που ασχολείται με τον πολιτισμό, λέμε ότι είναι μια γυναίκα που ασχολείται με τον πολιτισμό. Όταν είναι άντρα αυτός που ασχολείται με τον πολιτισμό, αρχίζουμε και βγάζουμε δεκάδες ονόματα. Μια τελευταία αυτοκριτική. Στα κείμενα που ετοιμάζουμε, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε εκφράσεις όπως οι γυναίκες ε, δεν υπάρχουν εκεί τιμητικά, ότι να είναι γυναίκες στα δυσυδικά συμβούλια γυναίκες που αποδεικνύουν, που είναι ικανές, που έχουν προσόντα. Πιστεύει κανείς ότι σε αυτό το επίπεδο θα δώσουν μια τέτοια θέση σε μια γυναίκα που δεν το αξίζει και υπεραξίζει, που δεν έχει αποδείξει την σταδιοδρομία της. Δείτε τα βιογραφικά των ευρωβουλευτών Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Να δείξουμε ταπεινοφροσύνη, να περάσουμε, αλλά να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλοί παντού και να έχουμε μία πρωτοπορία. Πρόκειται για δρόμο, για πορεία. Δεν θα σταματήσει. Ε, είναι ένας δρόμος για το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε μία συνέπεια στις πολιτικές μας. Αλλιώς ουδέποτε θα κάνουμε κάτι ουσιαστικό και να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση και τη δουλειά της κυρίας Κράτσα. Ελπίζω στο μέλλον να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε όλους αυτούς τους τομείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπιλμπάου. Κυρία Γκουρμά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Ρόδη Κράτσα για την έκθεση αυτή, γιατί είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι εμείς, οι γυναίκες, έχουμε ένα πολύ έντονο κόμπλεξ κατωτερότητας και ακόμα πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε όσο οι άντρες. Συζητάμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε θέση να καλύψουμε διευθυντικέ θέσει, Μα γιατί το συζητάμε καν αυτό αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο δεν διερωτώμαστε αν οι ίδιοι άντρε είναι ικανοί να καλύψουν τι θέσει αυτέ. Για ποιο λόγο να μιλήσουμε για ποσοστώσει για του ίδιου του άντρε. Για ποιο λόγο μιλάμε πάντα για ποσοστώσει σε σχέση με τι γυναίκε. Αν δεν είμαστε οι ίδιε σίγουρε για τη δικιά μα την αξία, αν δεν έχουμε ίδιε αρκετή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, δεν πρόκειται να σημειώσουμε πρόοδο. Η Ρόδη διάβασε όλες τις σχετικές μελέτες και κατέληξε σε κάποιες παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες ε, αν μία επιχείρηση, μία οργάνωση μπορούσε να έχει σε ηγετική θέση γυναίκες, θα κατέληγε να είναι και πιο αποτελεσματική. Και δυστυχώς οι άντρες δεν αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό. Για ποιο λόγο η Σουηδία αποφάσισε να εισάγει μία ποσόστοση για τις γυναίκες όσον αφορά τις ε, διευθυντικές θέσεις. Μα το κάναν αυτό επειδή ουσιαστικά να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να χάσουν την προστιθέμενη αυτή αξία που φέρνουν οι γυναίκες στις διευθυντικές θέσεις. Και βλέπετε ότι η χώρα αυτή έχει 40% και αναφέρομαι στην Νορβηγία αυτή τη στιγμή. Έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο του 40%. και αυτό έχει μεταφραστεί σε επιπλέον κέρδη για τις επιχειρήσεις αυτές. Υπάρχουν πλέον μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν σαφέστατα ότι επιχειρήσεις που απασχολούν υψηλότερο ποσοστό γυναικών στις διευθυντικές θέσεις είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν πολύ πιο εύκολα την οικονομική αυτή κρίση και πολύ πιο αποτελεσματικά δεν πρόκειται απλώ για μια θεωρητική προστιθέμενη αξία, πρόκειται για μια επιπλέον γνώση και εμπειρογνωμοσύνη που έρχεται με τι γυναίκε. ακόμα και αν δούμε και το επίπεδο εκπαίδευση και κατάρτιση. Ζήτημα το οποίο έθιξαν πολλοί συνάδελφοι άλλωστε και πάλι στο επίπεδο αυτό οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στα πανεπιστήμια. Το 60% των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες. Είμαστε λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν τα περισσότερα προσόντα και δυστυχώς χρειάζεται να συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εξίσου καλά με τους άντρες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το περίφημο γυάλινο πλαφόν για τις γυναίκες, πράγμα το οποίο δεν εφίσταται για τους άντρες. Η Επίτροπος Βίβια Ρέντινγκ μας είπε ότι αν εισάγουμε ποσοστώσεις τότε θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Ας δούμε όμως και τα στατιστικά δεδομένα για τελευταία δεκαέτη. Όσον αφορά την οικονομία πάντα. Κάθε φορά που μία γυναίκα καλύπτει μία διευθυντική θέση, μάλλον δεν έχει σημειωθεί ακόμα πρόοδος όσον αφορά το ζήτημα αυτό, την κάλυψη διευθυντικών θέσεων από τις γυναίκες. Τα στατιστικά δεδομένα δεν δείχνουν να έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Τουλάχιστον όμως σε πέντε κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι η κάλυψη διευθυντικών θέσεων από τις γυναίκες έχει οδηγήσει σε επιπλέον κέρδη, έχει οδηγήσει σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Δεν νομίζω πάντως ότι το παράδειγμα αυτό έχει ακολουθηθεί από πολλές χώρες και ότι δεν ακολουθούνται τα μέτρα αυτά αύξηση αποτελεσματικότητας από τις περισσότερες χώρες. Στις περισσότερες κοινωνίες τώρα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι ένα 52% των πολιτών είναι γυναίκες, το 48% είναι άντρες. Ο ο Γιώ Λάινεν είπε ότι θα πρέπει και προς αυτό να υπάρχουν ποσοστώσεις. Η πρωτοβουλία όμως αυτή απέτυχε. Δεν καταφέραμε να αυξήσουμε την συμμετοχή των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό που βλέπουμε στην υφιστάμενη οικονομική κρίση είναι ότι οι πρώτες θέσεις οι οποίες καταργούνται, οι πρώτες θέσεις εργασίας που καταργούνται είναι οι θέσεις των γυναικών. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό και αποσαφήνισαν ότι το ζήτημα δεν είναι να μας αρέσουν οι ποσοστώσεις ή όχι, είναι τελικά η αναγνώριση ότι οι ποσοστώσεις είναι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο που έχουμε στη θέση μας αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ο Μπαρόσο συνέστησε την πρώτη του Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρώτη ομάδα έλαβε ιδιαίτερα υπόψη την εκπροσώπηση των γυναικών. Στη δεύτερη όμως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε κάτι τέτοιο. Μόνο τρεις γυναίκες τελικά διορίστηκαν από τα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια ο Μπαρός άρχισε να στέλνει διάφορα μηνύματα στα κράτη-μέλη λέγοντας ότι αν στείλετε γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε είναι πιο πιθανό για αυτήν να τη ανατεθεί ένα χαρτοφυλάκιο πιο σημαίνον, μπορούμε να πούμε, πιο σημαντικό. Και είδαμε ότι υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη που εξαιτία αυτού του επιχειρήματο αποφάσισαν να μην διορίσουν γυναίκες υποψηφίους. Εμείς επίσης είπαμε ότι δεν συμφωνούσαμε το γεγονός ότι τελικά θα είχαμε τρεις γυναίκες μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κινητοποιήσαμε λοιπόν ε, εκ νέου τα κράτη-μέλη προκειμένου να αλλάξει αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που είπα στην αρχή. Χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί χωρί τα χαρακτηριστικά αυτά δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου μα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Γκουρμάη. Η κυρία Πλάμ έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλα αυτά τα οποία έκανε και έγραψε στην έκθεση αυτή η συνάδελφός μας Ρόδη Κράτσα. Συμφωνώ με την χρησιμοποίηση του σημαντικότατου αυτού πολιτικού μέσου. Πρόκειται για ένα πολιτικό, ρεαλιστικό μέσο το οποίο το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ επίσης με τους προλαλήσαντες. Πέρα από το μηχανισμό των ποσοστώσεων χρειαζόμαστε και κάποια συμπληρωματικά μέτρα. Αναφερόμαστε στην άδεια μητρότητα, στην άδεια πατρότητας, γονική άδεια και όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Και να σα πω κάτι ακόμα. Έρχομαι από τη Ρουμανία και στην χώρα μου ακούμε πολύ συχνά και το άκουσαν το λέει και η ίδια η Vivian Redding ότι ε, χρειαζόμαστε ίση μεταχείριση σε όλο το φάσμα των κοινωνιών παντού στην Ευρώπη. Πρέπει να μιλάμε όλο και περισσότερο για τη διάσταση των φύλων παντού στην κοινωνία μας. Οι γυναίκες στη Ρουμανία όταν άκουσαν την δήλωση της Vivian Redding σχετικά με τις ποσοστώσεις και ότι θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τις επιχειρηματικές ηγετικέ θέσεις, αναρωτήθηκαν «Μα τι θα γίνει με την πολιτική» Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται μία ανάλογη πρωτοβουλία για τον πολιτικό τομέα. Και όπως, όπως είπε η Μπάρμπαρα πριν από λίγο, στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλα κρατημέλα, ακόμα και στη Ρουμανία, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται. και οι γυναίκες θα ήθελαν να εισαχθούν και στις περιπτώσεις αυτές ποσοστώσεις. Αρκεί όμως οι ποσοστώσεις αυτές να είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Αν όμως οι ποσοστώσεις ισχύουν μόνο για τις επιχειρηματικές ηγετικές θέσεις, τότε θεωρούν ότι γίνεται πάλι μία διάκριση. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή γυναικών σε μία επιχείρηση. Όσο περισσότερες είναι οι γυναίκες στις επιχειρηματικές ηγετικές θέσεις, τόσο αυξάνεται και η προστιθέμενη αξία για την ίδια την επιχείρηση. Υπάρχουν όμως ανάλογες μελέτες που να αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρουν οι γυναίκες στην πολιτική. Και υπάρχουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και θα πρέπει να σταλεί ένα πολύ ηχηρό μήνυμα και πρέπει να το στείλουμε εμεί ω το πιο δημοκρατικό θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά την ε, εισαγωγή τέτοιων πολιτικών μέσων προκειμένου να διορθώσουμε την κατάσταση και να αυξήσουμε την εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τομείς σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας. Γιατί πραγματικά πρέπει να καταλήξουμε τελικά σε μια πλήρως δημοκρατική κοινωνία. Και έχουμε ήδη δει ότι στα κράτη-μέλη εκείνα που υπάρχει ίση εκπροσώπηση αντρών και γυναικών, υπάρχει και ίση μεταχείριση και στις κοινωνίες τελικά αυτές βλέπουμε ότι η πρόοδος είναι πιο γρήγορη, η δημοκρατία είναι πολύ πιο ισχυρή και η εκπροσώπηση είναι πολύ πιο ισορροπημένη σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Υποστηρίζω πλήρως τα όσα είπαν οι συναδελφοί μου και συμφωνώ απόλυτα με την παρουσίαση της κυρίας Κράτσα. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ακόλουθο να αρχίσει να σκέφτεται λίγο ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την ίση μεταχείριση παντού στην κοινωνία. Ευχαριστώ. η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σχεδόν τα είπαμε όλα, αλλά το γεγονός ότι το, ότι το συζητάμε τόσο πολύ και όλοι σχεδόν μίλησαν και όλο και περισσότερες αποδείξεις του προφανούς κομίζουμε, δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε να εντοπίσουμε αυτές τις διακρίσεις. Διακρίσεις είναι αυτές. Μιλάμε για καλά εδρεωμένες ιστορικές διακρίσεις και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την έκθεση στην κυρία Κράτσα. Δεν θα είναι εύκολο, δεν είναι μόνο οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις κλπ. κλπ. Αν δείτε πώς κάποια κράτη-μέλη δεν αξιολογούν ούτε τα θέματα της άδεια μητρότητα. Είναι ακόμα απρόθυμα να αναγνωρίσουν την πλήρη αμοιβή κατά τη διάρκεια της άδεια μητρότητα. Θεωρούν ότι αυτό είναι ίσονο σημασία για την κοινωνία. Ενώ πώς θα αναπαραχθεί η κοινωνία με τα παιδιά που γεννούν οι γυναίκες και όμως το υπονομεύουν αυτό. Επίσης, δείτε πόσες εκθέσεις υπάρχουν για αυτό το θέμα κανείς δεν θέτει το ερώτημα γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή τη δημοσιονομική χρηματοοικονομική κρίση. Ποια ήταν η ευθύνη των γυναικών. Υπάρχουν τρεις μελέτες της Deutsche Bank, McKenzie κλπ. Και αποδεικνύουν ότι οι χώρες και οι εταιρείε που ε, είχαν επικεφαλής γυναίκες ως top manager ή είχαν γυναίκα πρόεδρο του Συμβουλίου, τα κατάφεραν μια χαρά. Κανείς όμως δεν ρωτάει ποιος δεν τα πήγε καλά και τι έγινε μετά, τι συνέπειες υπήρξαν. Όταν μιλάμε για ποσοστώσεις, απογοητεύομαι πολύ όταν ακούω κάποιες γυναίκες να λένε δεν θέλω να πάρω τη θέση μιας υψηλής θέσης μόνο επειδή είμαι γυναίκα και επειδή υπάρχει ποσόστοση. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτή είναι παρερμηνία. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να μας εξοβελήσουν επειδή είμαστε γυναίκες. Προλαμβάνει το μέτρο αυτό την περιθωριοποίηση και τη διάκριση. Δεν ισχύει το αντίθετο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις ποσοστώσεις. Και όπως είπε και η Μαρή Κορνέλισεν, εμείς βελτιώνόμαστε κατά μισό τα εκατό ετησίως. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Και όλα τα μέτρα, όλα τα βήματα θα ληφθούν κατά της κατάστασης. Κάποια στιγμή μπορεί να θεσπιστεί βραβείο Ζαχάροφ εδώ στο Κοινοβούλιο για κάποιον που προασπίζεται όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αφρική, αλλά για την προάσπιση των ε, δικαιωμάτων των γυναικών εδώ, στην Ευρώπη, που είναι γελίο, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε η καλύτερη δημοκρατία και το καλύτερο παράδειγμα παγκοσμίωση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ γενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτή λοιπόν είναι μια παράδοξη συζήτηση και το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί στο, στην Προεδρία. Εδώ η συνάδελφος Μπιλμπάου μίλησε για τις προεδρίες, μίλησε για την ανδροκρατούμενη εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση στα αξιώματα. Πόσο θα το ανεχθούμε αυτό, πόσες συζητήσεις χρειάζονται ακόμα, πόσες φορές πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε, πόσες εκθέσεις ακόμα θα πρέπει να καταρτήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι ξεκάθαρο πια. Και τέλος, ιστορικά υπάρχουν εδρεωμένες διακρίσεις και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές γιατί είναι ντροπή. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους για την ωραία συζήτηση, την ενδιαφέρουσα, την έντονη εντατική και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που συμμετέσχουν και αποδεικνύουν πόσο αφοσιωμένοι είναι στο θέμα αυτό. Δίνω το λόγο τώρα στο Ιρώδη Κράσα για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που έχουν για την έκθεση και τον κοινό στόχο που θέλουμε να υπηρετήσουμε να είναι το μήνυμά μας σαφές και καθαρό. Και ε, δόθηκε ευκαιρία να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση και για θέματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την έκθεση και φαίνεται πραγματικά αυτό που είπε η κυρία Παρβάνοβα μόλις ότι τόσες εκθέσεις που έχουμε κάνει, τόσες φορές που έχουμε ασχοληθεί με τα γενικά θέματα γυναίκες στην πολιτική, γυναίκες στην εργασία, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, πόσο αυτά τα θέματα αισθανόμαστε ότι πρέπει με κάθε ευκαιρία να τονίζονται και με την ευκαιρία επιτρέψτε μου προτού φτάσω στο θέμα το συγκεκριμένο της δικής μου έκθεση ότι θα πρέπει να προσγειωθούμε στην έκθεση που συζητούμε ε, αφιερώνουμε κάθε χρόνο την 8η Μαρτίου στο θέμα γυναίκες και πολιτική. Κάνουμε και μια μεγάλη εκδήλωση στο Κοινοβούλιο με, την ε, ευθύνη της Επιτροπής μας ε, και προσκαλούμε αντίστοιχες επιτροπές από τα εθνικά κοινοβούλια. Έχω την αίσθηση, κυρία Πρόεδρε και αγαπητέ συνάδελφοι, ότι δεν έχουμε ούτε προβάλλει επαρκώς ούτε αξιοποιήσει το γεγονός αυτό. Το λέω επειδή το να αποφασίζουμε κάθε χρόνο να κάνουμε αυτή την, ε, αυτή την εκδήλωση σημαίνει ότι είναι για μας ένα μείζον θέμα που το συνδέουμε απόλυτα με την 8η Μαρτίου παράλληλα με τα άλλα γεγονότα που κάνει το Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι και η... καταρχάς δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή ως φορές έρχομαι, πηγαίνω στην εκδήλωση αυτή, μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη μας ε, αλλά ούτω ή άλλω πιστεύω είχα σκοπό να το ζητήσω και η σημερινή συζήτηση μου δίνει την ευκαιρία να γίνει μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων να τα διαδώσουμε αυτά να κάνουμε ένα follow up. δεν ε, ε, αρμόζει σε ένα τέτοιο στόχο να τον ανακαλύπτουμε και να τον συζητούμε κάθε 8η Μαρτίου. Ε, πανέρχομαι τώρα στην έκθεση. Ήταν πολύ γενικά και πολλά συγκεκριμένα αυτά τα οποία τέθηκαν. Ε, Πιάνω τα συγκεκριμένα μόνο, γιατί αυτά θα συνδεθούν με την έκθεση περισσότερο. Ε, ήθελα να απαντήσω στην κυρία Κορνέλισεν, η οποία έχει μια συνεχή παρουσία και συμμετοχή ε, πρώτον απορώ για την εντύπωση που της δόθηκε ότι δεν ήταν ε, συνεργάσιμη το κλίμα στην ε, ε, συνάντηση που κάναμε για, τα, για τις διαπραγματεύσεις, για, το, για να φτάσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. δεν έχουν την ίδια εντύπωση άλλοι συνάδελφοι και ίσως κάποια παρεξήγηση, κάτι δεν καταλάβατε καλά. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν εκφράζει εμένα η μη διάθεση συνεργασία. Συγκεκριμένα σε αυτό που είπατε για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την ανάγκη απειλών. Ε, η έκθεση το κάνει σαφές. Φυσικά η λέξη απειλέ, δεν είναι μια λέξη η οποία μπορεί να μπει, ε, χαιρετίζουμε τι απειλέ, να μπει σε ένα σε μια παράγραφο αλλά εν πάση περιπτώσει χαιρετίζει τα μέτρα της επιτροπής η έκθεση και τονίζει αν διαβάσατε καλά και την αιτιολογική έκθεση και τα, και τα, α, λαμβάνοντας υπόψη ότι και μόνον τονίζω και μόνον ο, στα, στις χώρες που εκφράζεται η πολιτική βούληση για νομοθετικά μέτρα και ποσοστώσεις αρχίζει κάποια εξέλιξη. Άρα γίνεται σαφές στην έκθεση ότι χρειάζεται αυτό το ταρακούνημα των νομοθετικών μέτρων. Ε, ήθελα να πω για τον κύριο Ταραμπέλα, ο οποίος αναφέρθηκε, λείπει ο κύριος Ταραμπέλα, αλλά το συγχωρούμε γιατί συνήθως είναι πολύ συνεπής, ε, αναφέρθηκε στις εμπειρίες από την Ορβηγία, από τη Γαλλία, από, μέτρα, από άλλες χώρες. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της πρώτης, συμβιβαστική ε, του της πρώτης πρότασης και επίσης κάναμε μια δημόσια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας με γυναίκες από την ε, Νορβηγία που είχαν ευθύνη της εφαρμογής του νόμου από τη Γαλλία, την εισηγήτρια του νόμου από τη Γαλλία και επίσης γυναίκες εκπροσώπους δικτύων διεθνών για να δούμε πώς είναι και η διεθνής εμπειρία αυτό να έχετε υπόψη σας για όσους δεν το παρακολουθήσατε ότι η Επιτροπή μας επένδυσε σε αυτό μετά από τη δική μου πρόταση και κάναμε αυτή τη δημόσια ακρόαση και ε, τονίσαμε και τιμήσαμε την εμπειρία που υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο και στο διεθνή χώρο ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στον κύριο Ρωμέβα, ο οποίος παρουσίασε αυτή όλη την προβληματική που υπάρχει στον χώρο της εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στην έκθεση αυτή δεν είναι το πλαίσιο, η έκθεση έχει συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όλη την ε, προβληματική της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Έχουμε κάνει άδειες ε, εκθέσεις, θα έχουμε στο μέλλον σίγουρα που θα αναπτυχθούν. Θέλω όμως να πω ότι ήδη αυτό αναφέρεται ε, στην έκθεση, ε, στο μέτρο που η έκθεση το επιτρέπει, ο χώρος και το θέμα, ότι πρέπει να διευκολυνθεί να μπορούν να εργαστούν ε, οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, χωρίς εμπόδια, χωρίς διακρίσεις. Και θέλω να σας πω κάτι κύριε Μέβα, ακόμη και εκεί που είναι γυναικοκρατούμενες επιχειρήσεις, που είναι αρνητικό για την παραγωγή και για την έκφραση των γυναικών, και εκεί που είναι γυναικοκρατούμενες επιχειρήσεις, ε, και τη ελαφρά βιομηχανία συνήθως και εκεί στα διοικητικά συμβούλια είναι άνδρες. Άρα δεν φταίει το ότι δεν είναι άνδρες εργαζόμενοι, φταίει η νοοτροπία ότι οι γυναίκες μπορεί να εργάζονται καλά, να κάνουν ραπτική, κοπτική, αλλά οι άνδρες θα διευθύνουν το management. Λοιπόν, δεν, συνδέονται απόλυτα οι γυναίκες εργαζόμενες και το management. Ε, θέλω επίσης να αναφερθώ στην... Ε, ε, στο αυτό που είπε ε, να κάνω ένα συνδυασμό με αυτό που έθεσε Ζήτα Γκουρμάη, ότι πέρα των συνθήκων που είναι δυσχερών για τις γυναίκες, είναι και έλλειψη φιλοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Και γι' αυτό, αυτό μου εντυπωσίασε στις μελέτες που είπε Ζήτα ότι διάβασα για να μπορέσω να καταλήξω κάπου, ότι οι παράμετροι, οι αρνητικές στο να φτάσει μια γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι δυσκολία συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Συνήθως οι γυναίκες που ξεκινάνε με εφόδια, που θέλουν να κάνουν μια καριέρα, που έχουν μια ανέλυξη, έχουν ένα καλό μισθό, ε, ε λύνουν το πρόβλημά τους αυτό, στο πλαίσιο που ένα πρόβλημα τέτοιο μπορεί να λυθεί. Είναι μετά ότι οι ίδιες δεν επενδύουν και επίσης δεν υπάρχουν τα μέτρα στην επιχείρηση. Γι' αυτό δίνω έμφαση στο mentoring, στο networking, στην ε, ε, παρακολούθηση της προσωπικής καριέρας μιας γυναίκας. Ε, δεν ξέρω για όσους έχετε ασχοληθεί και έχετε παρακολουθήσει, υπάρχουν τέτοια προγράμματα, αλλού είναι επιτυχημένα, πιο πολύ, αλλού λιγότερο, που είναι αντικείμενο μια γυναικεία καριέρα που δηλώνει ότι θέλω να φτάσω κάπου, έχει μια, ενα ένα follow-up. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η, έλλειψη παιδικών σταθμών που τονίζω αυτό. Παίρνω και τη κυρία Ματέρα και άλλων την, ε, μέσα την, ε, και τη κυρία Κώστα ότι πρέπει να υπάρχουν και φορολογικέ ε, κίνητρα, φορολογικά κίνητρα, να δημιουργηθούν παιδικοί σταθμοί, άλλες facilities κτλ. Αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Θέλει πα, ε, πολλούς παράγοντες μαζί για να φτάσει μια γυναίκα σε ένα διοικητικό συμβούλιο θέλει και την προσωπική της επένδυση και θέλει να αισθανθεί ότι μπορεί πέρα από το να αφήσει κάπου το παιδί της ή να τη διευκολύνει ο σύζυγος πρέπει να υπάρχει και μέσα στην επιχείρηση μια, ένα mentoring και μια αντιμετώπιση θετική. Γι' αυτό δίνω έμφαση στην ευθύνη και την ευαισθητοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη πλευρά θέλω να σας πω ότι αυτό το καινούριο που μου βγήκε σήμερα από τη συζήτηση που κάναμε διότι μερικά πράγματα επαναλαμβάνω πάντα στο, θέμα της έκθεσης διότι ακούστηκαν πράγματα που άγγιξαν τις ψυχές μας και θα δοθούν ευκαιρία να κάνουμε καμπάνιες όπως είναι το θέμα του, της εκπροσώπησης των το... το γυναικών στις... στις θέσεις απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό και εν ώψη των ευρωεκλογών που έρχονται και των άλλων θεσμικών οργάνων. Μπορούμε να κάνουμε μια καμπάνια, να πάρουμε το 50-50 που είχε ξεκινήσει την περασμένη φορά, να κάνουμε μια καμπάνια πιο όρημη, πιο απαιτητική, πιο συγκεκριμένη και πιο διαδεδομένη σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες. Γιατί δεν έχει φτάσει το μήνυμα την περασμένη φορά σε όλες τις χώρες, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι χώρες εκφράζουν το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης τα πολιτικά κόμματα. Διότι τα πολιτικά κόμματα αποφασίζουν για το πώς μοιράζονται οι θέσεις εδώ, ποιους προτείνουν προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέδρους των πολιτικών ομάδων. Λοιπόν, θα έχουμε τέτοια ευκαιρία. Επανέρχομαι, προσγειώνομαι στην έκθεση τη σημερινή. Αυτό που ε, νομίζω ότι μπορούμε να τονίσουμε περισσότερο και θα κάνω μια πρόταση είναι η ανάγκη ευαισθητοποίησης. Ε, πήρα την, ε, την ιδέα από συναδέλφους και έχω μια παράγραφο για τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Διότι πρέπει και οι κοινωνικοί εταίροι να ευαισθητοποιηθούν. Είτε οι σύλλογοι επιχειρήσεων, τα επιμελητήρια, τα συνδικάτα να ενημερωθούν για αυτή την αξία, την ηθική και την οικονομική της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Χρειάζεται όμως μια ευρύτερη καμπάνια ευαισθητοποίησης. Διότι και η κοινή γνώμη πρέπει να καταλάβει αυτή τη σημασία. Και επίσης προς την κυρία Κώστα, την οποία ευχαριστώ για όλη την ε, καλή διάθεση συνεργασίας, θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό που τόνισε η κυρία Κώστα, καμιά φορά και η διερμηνία δεν μας βοηθά να καταλάβουμε κάποιες πτυχές, όσο και αν οι διερμηνείς κάνουν εξαιρετική εργασία, μόνιμα, χωρίς αυτές και αυτούς δεν μπορούσαμε να υπάρξουμε. Ε, αναφερθήκατε στο θέμα της αξιολόγησης, της αξιοκρατίας, των βιογραφικών θέλω εδώ αν μου επιτρέψετε κυρία πρόεδρε να κάνω μια, ε, μια ε, έτσι, παρέμβαση ιδιαίτερη. κοιτάξτε η επιχείρηση δεν είναι γραφειοκρατία. η επιχείρηση επιμένει ότι θέλει ότι σε, έναν, σε μια γυναίκα που θα, και έναν άνθρωπο που θα της ε, αναθέσει μια θέση ευθύνη του management ψάχνει και άλλα στοιχεία. Ε, μπορεί να υπάρξει ένα πολύ καλό βιογραφικό το βλέπουμε και εμείς όταν βλέπουμε, ε, ψάχνουμε ε, βοηθούς ένα καλό βιογραφικό που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που χρειάζεται στην ευελιξία στην ετοιμότητα στο feeling της αγοράς δηλαδή δίνω μεγάλη έμφαση στην αξιοκρατία και στην διαφάνεια και στα skills όπως τα έχουμε βάλει σε διάφορες συμβιβαστικές παραγράφους αλλά να ξέρετε ότι ε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ έχω αυτό το βιογραφικό και δεν με προάγαγαν σε αυτή τη θέση όπως μπορεί να το διεκδικήσει σε μια administration, σε public administration. Λοιπόν, εκεί οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη του αποτελέσματό τους και ψάχνουν τους κατάλληλους. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για το κινητικό honorary position στην οποία αναφερθήκατε. Καταρχάς η λέξη αυτή έχει φύγει διότι δημιουργεί διάφορες παρεξηγήσεις και υπάρχει μια συμβατιστική τροπολογία που αναφέρεται σε αυτό που ήθελα να πω, αλλά δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Δεν καταλάβατε καλά το πνεύμα. Θέλω να πω ότι όταν πιέσουμε πολλές επιχειρήσεις, ήδη υπάρχουν κάποια τέτοια περιστατικά στη Γαλλία, ας πούμε, πιέσουμε επιχειρήσεις. Κυρίως επιχειρήσεις που είναι σε μορφή οικογενειακών επιχειρήσεων, τις πιέσουμε για να βάλουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, θα πούνε εύκολα είναι η κόρη μου, η γυναίκα μου, έχουν πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις, η κόρη μου έχει πάρει ένα πτυχίο, είναι άξια για το διοικητικό συμβούλιο. Η γυναίκα μου έχει εμπειρία 20 χρόνων που εργάζεται εδώ, είναι άξια για το διοικητικό συμβούλιο. Η ανιψιά μου κτλ. Αυτό ήταν το θέμα, ότι ο στόχος, αν δείτε τη συμβαστική τροπολογία όπως είναι γραμμένη, όχι την αρχική, τη συμβαστική. Είναι η τροπολογία 2 λέει ότι ο στόχος του να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια δεν πρέπει να βασίζεται ε, σε θέσεις που δίνονται έτσι για να αυξηθεί ο αριθμός αλλά σε γυναίκες που έχουν τα προσόντα διότι εμείς ξέρουμε, φάνηκε και σήμερα πόσο υποστηρίχθηκε από εδώ ότι υπάρχουν γυναίκες που τα έχουν γυναίκες που έχουν κάνει καριέρα μέσα στην επιχείρηση ή σε κάποιες θέσεις γυναίκες που έχουν μια ειδικότητα από ένα χώρο. Αυτό ήταν το πνεύμα, να μην είναι μια γυναίκα ε, του φιλικού, του, του, του, ή ε, που εξυπηρετεί κάποιες δημόσιες σχέσεις ε, και δεν είναι μια γυναίκα που αξίζει να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι ε, μπορούμε να, έτσι, να τονίσουμε αυτά τα θέματα τα οποία μας βρίσκουν όλους και όλες ε, σύμφωνους και το, ε, κατά την άποψή μου αυτό που εγώ θα κάνω μια πρόταση είναι να τονιστεί εκεί που λέμε για το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους να βάλουμε και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και, των, και της κοινή γνώμης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε κυρία Κράτσα. Θα ψηφίσουμε στις 25 Μαΐου στην Επιτροπή και μετά θα πάρει το δρόμο για την Ολομέλεια τον Ιούλιο η έκθεση. Πριν πάμε στο επόμενο σημείο, στην ημερήσια διάταξη, θέλω να ρωτήσω όλους τους συναδέλφους να είναι όσο γίνεται πιο σύντομοι όταν ζητούν το λόγο, γιατί έχουμε άλλα πέντε σημεία στην ημερήσια διάταξη και η συζήτηση σήμερα για αυτό το θέμα κράτησε μία ώρα και ένα τέταρτο. Αυτό το θέμα πήγαινε για ψηφοφορία και μας πήρε τόσο χρόνο. Να είστε σύντομοι λοιπόν. Έχουμε 15 λεπτά για κάθε θέμα από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να προλάβουμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης για την Επιτροπή Προϋπολογισμών, εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012. Η κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα είναι η ε, υπεύθυνη εδώ. Να πω ότι όταν το κυκλοφόρησε το σχέδιο γνωμοδότησης δεν είχαμε πρόσβαση στις συγκεκριμένες προτάσεις από την Κομισιόν. Τώρα όμως έχουμε πρόσβαση. Άρα τροποποιήσαμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ώστε να μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις που ήρθαν και από την Κομισιόν. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη κυρία Πρόεδρε. Τον Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2010-2015 και επανεπιβεβαίωσαν πόσο σημαντικό είναι να δοθεί μάχη για την ισότητα των γυναικών στον χώρο εργασίας. Και αυτό χρειάζεται και στο, στην, στην πολιτική αρένα, όπως είδαμε σήμερα, και χρειάζεται περισσότερη ισότητα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, όπου ένας στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων. Άρα περισσότερη ισότητα επιδιώκεται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει τον στόχο την αύξηση, ως στόχο την αύξηση της ισότητας και της απασχόλησης των γυναικών. Έχουμε 62% ε, τώρα και η στρατηγική θέλει ποσοστό απασχόλησης γυναικών 75%. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσβλέπει στη μεγέθυνση βιώσιμη μεγέθυνση ανάπτυξη στην οικονομία και για να επιτευχθούν αυτές, αυτοί οι στόχοι χρειαζόμαστε περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, μεγαλύτερη υποστήριξη στις γυναίκες, γυναίκες από ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, πιο ηλικιωμένες, μόνες γυναίκες, μονογονικές οικογένειες, γυναίκες με αναπηρία, μετανάστριες. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης εξέτασα κυρίως την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βίλνιους για την ισότητα των φύλων, διότι ε, κάνουν έρευνες οι οποίες δίνουν πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις προσλήψεις προσωπικού. Υπάρχει πιλωτικό έργο που εξετάζει την, ε, στον συνδυασμό της ε, ζωής στην εργασία και στην οικογένεια για τις γυναίκες. Και κάτι άλλα πιλωτικά έργα εξετάζουν και καινούργια θέματα που θα μας απασχολήσουν στην Επιτροπή. Την κατάσταση των, γυναικών, των μόνων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση των γυναικών στο ζήτημα αυτό ο αριθμός των single mothers στην Ευρώπη αυξάνεται εκθετικά και οι δυσκολίες ε, υπάγονται σχετίζονται με τον αποκλεισμό και την κοινωνική κατάσταση των ίδιων και των παιδιών τους. Ελπίζω να πηγαίνω αρκετά γρήγορα, υπερβολικά γρήγορα για τους Γερμινείς. Για το draft opinion τώρα εδώ, περιορίστηκα και στην ανάγκη να μειωθούν οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην κατάσταση των ηλικιωμένων που είναι περισσότερο ευάλωτες και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και τις φτωχές γυναίκες, ιδίω υπό το φως του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργή γύρανση, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε πόρους για, την, ε, για το κόστος κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης όπως είπε και η πρόεδρο, προσπαθώ να τελειώσω γρήγορα. Παρουσίασα την έκθεση αυτή χωρί να έχω ένα feedback ε, του σχεδίου προπολογισμού 2012 της Επιτροπή που, θα που υποβλήθηκε σήμερα το πρωί. Θα δω λίγο χρόνο για να υποβάλω και τροπολογίε λοιπόν με βάση το κείμενο αυτό. Ζητώ από του συναδέλφου να μου στείλουν όσο περισσότερε τροπολογίε ε, θεωρούν. Ευχαριστώ. Και εγώ. Ευχαριστούμε κυρία Ματέρα. Κύριε Γκουρμά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη. Τονίσατε κάποια πολύ σημαντικά θέματα κύριε Ματέρα. Η στρατηγική για την ισότητα δεν περιλαμβάνει την εργασιακή διάσταση. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε σημασία στην σπουδαιότητα των πιλωτικών έργων στον τομέα αυτό. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη την κατάσταση των ε, ανήπαντων μητέρων, των μητέρων μόνων. Είμαι σκιωδησυγήτρια για το ζήτημα αυτό και είμαι βέβαιο ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της μισθολογικής ε, απόκλησης. Είμαι πεπισμένο ότι το νέο σύμφωνο που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 8 Φεβρουαρίου αποτελεί ένα βήμα μπρος. Να σας πω απλά ότι μεταξύ 2006 και 10 Υπήρχε, υπήρξε επίσης ένα σύμφωνο ισότητα, όπου επίσης γίνονταν προσπάθεια να υπερκεραστεί η μισθολογική ανισότητα, αλλά δεν είδαμε πολύ πρόοδο. Η κυρία Μπάουρ ετοίμασε μια εξαιρετική έκθεση σχετικά στην προηγούμενη θητεία. Αν όμως δεν υπάρξει μια ε, οδηγία για τη μισθολογική ανισότητα, δεν θα αλλάξει η κατάσταση των γυναικών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει σχετική μνήμα. Μία διευκρίνηση. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά, αλλά η στρατηγική για το φύλλο ενώπιση του 2000, στην στρατηγική του 2020 είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη. Πρέπει να υπάρξει ισότητα στην αγορά εργασία, αλλά δεν μιλάνε για στατιστικά στοιχεία. αύξηση των, ε, της απασχόλησης από 50-60% στις γυναίκες και από 60-70% στους άνδρες. Αλλά μόνο αυτά τα νούμερα υπάρχουν. Άλλα νούμερα δεν βλέπω να υπάρχουν. Καλό θα ήταν λοιπόν να μιλούμε για στοιχεία. Να μιλήσω για την κατάσταση των ηλικιωμένων. Δεν είναι μόνο ευάλωτες οι μόνες γυναίκες αλλά και οι ηλικιωμένες. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μογασαντιέ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητάμε αυτή τη στιγμή την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προπολογισμού 2012. Θα ήθελα λοιπόν να, να κάνω μια πολύ απλή συγκεκριμένη παρατήρηση που ουσιαστικά συνάδει μετά όσα είπε και η κυρία Γκουρμάη. Θα θέλαμε να συγκλίνουν περισσότερο οι πολιτικές προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών. Θα ήθελα λοιπόν στην εντολή αυτή τη διαπραγματευτική να έχουμε μία πραγματική, ξεκάθαρη δημοσιονομική παρουσίαση των πόρων που θα δοθούν για την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, ποιο θα είναι το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, αναφερόμαστε στο πρόγραμμα Progress, στο κοινωνικό ταμείο, το πρόγραμμα Δάφνη κατά της, των διοτήτων. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε συνεπείς, πιστεύω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε προκειμένου τα κοινωνικά αυτά ταμεία τα οποία σχετίζονται με τις συγκεκριμένες αυτές πολιτικές να είναι πιο ξεκάθαρα ως προς τη χρηματοδότησή τους. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα και δεν έχουμε και καμία φιλοδοξία. Σας ευχαριστούμε η κυρία Φιγκερέρου. Εκτός μικροφόνου. Ε, Ήθελα να κάνω τρία σχόλια σημαντικά. Πρώτον, με το αφορούν τον ε, χώρο της εργασίας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται πόροι όπως το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ενίσχυση της έμφυλης ισότητας, ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας. Εξίσου σημαντικό ωστόσο είναι αυτό το οποίο απαξιώνεται γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, δεν υπήρξε μια σωστή απάντηση όπως το Equal για παράδειγμα, πρέπει να το λάβει υπόψη η Επιτροπή. Έχουμε το Progress με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Δόθηκαν πόροι για την δημιουργία νέων πρωτοβουλειών. Αυτό οδήγησε σε ανεπαρκή χρηματοδότηση. Άρα πρέπει να επιμείνουμε στην Επιτροπή να χρηματοδοτήσει με κατάλληλο τρόπο το πρόγκρες. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι βιώνουμε σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης. Πολλές φορές είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν συμμετοχή 20% όπως απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης δεν υποβάλλονται έργα διότι δεν υπάρχει το 20% για την ε, συμμετοχή που απαιτείται. Σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως η Πορτογαλία αυτό είναι το ήθη, το σύνηθες. Πρέπει λοιπόν να πούμε στην Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Στο παρελθόν η κατάσταση δεν ήταν τόσο κακή και είχαμε και πετυχαίνουμε που και που να φτάσει το 10% η συμμετοχή αυτή. Καλό θα ήταν να επανέλθει και τώρα η Επιτροπή στο ποσοστό αυτό, την συμμετοχή 10, με, με, με ίδια κεφάλαια 10% των οργανισμών κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί αλλιώ χάνουμε τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε έργα που χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά όργανα διότι οι κοινωνικοί οργανισμοί δεν έχουν, αυτές οι κοινωνικές οργανώσεις δεν έχουν το αναγκαίο κεφάλαιο. Καλύτερα λοιπόν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά κονδύλια αν δίναμε έμφαση σε αυτή τη διάσταση. Καλά τα λόγια, αλλά μετά φράγκα δεν υπάρχουν για να υλοποιηθούν. Θα υποβάλω απολογίες για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω αυτά τα ζητήματα προς όρους συναδέλφου. Σας ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Η κυρία Ματέρα θα πάρει το λόγο για να συνοψίσει την όλη συζήτηση. Να ευχαριστήσω όμως πρώτα όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια γιατί πραγματικά καταβάλατε πολύ σημαντική προσπάθεια προκειμένου να είστε σύντομοι. Κύριε Ματέρα, έχετε το λόγο. Όχι, δεν θέλω. Κάνω σχόλια σε αυτά που μου είπαν οι συνάδελφοι. Διότι στην ουσία αυτό που θύμος, θύμισαν είναι σημαντικό. Το πιστεύω κι εγώ. Ιδίω αυτά που είπε η κυρία Φιγκερέδο στην παρέμβασή στην την δυνατότητα να μειώσουμε τη συγχρηματοδότηση στο 10%. Διότι πολλά κρατημέλη και όχι μόνο στου τομείς αυτούς χάνονται έργα λόγω τη αδυναμία συγχρηματοδότηση. Περιμένω τι τροπολογίε, θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσω να βελτιώσουμε την καλύτερη opinion που θα μπορέσει να παρουσιάσει η Επιτροπή στο μέλλον. Eh, ευχαριστούμε κυρία Ματέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν υπάρχει πρόσωπος ευρωπαϊκή επιτροπή σήμερα για να μας μιλήσει για, την, για το ζήτημα αυτό. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 3 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στι 25 Μαΐου. Και θα πάει στην Επιτροπή Προπολογισμών αυτή γνωμοδότηση 14 Ιουλίου και στην Ολομέλεια στην δεύτερη ολομέλεια του Ιουλίου. Του, του Ιουνίου, Στη συνέχεια έχουμε μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη των ατόμων αναπηρίες και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απηρία 2010-2020. Υπεύθυνη για την Επιτροπή μας είναι η Αντιπρόεδρός μας, κυρία Μογάν Σαχτιέ. Της δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω το όλο πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πρότεινε ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στους, στις σημαντικότερες αρχές, σημαντικότερους στόχους της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στα κράτη-μέρη. Η βασική λοιπόν έκθεση είναι η έκθεση ΚΟΖΑ στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πολύ, πολύ προσεκτικά λοιπόν διάβασα τις προτάσεις που γίνονται εκεί προτάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα συνεκτικές. Με συγχωρείτε, λέει η ομιλήτρια. Προτάσεις λοιπόν οι οποίες συνάδουν ιδιαίτερα με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας πω ότι για την γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε εμείς ως Επιτροπή προτείνω μία προσέγγιση πολύ συγκεκριμένη, πολύ πραγματιστική που αναφέρεται κυρίως στις δικές μας αρμοδιότητες και ευθύνες. Αυτές δηλαδή που έχουμε στα πλαίσια της δικής μας της Επιτροπής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα πρώτα δύο σημεία επί των οποίων πιστεύω ότι θα πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας είναι η κοινωνική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατομμυρίων ατόμων με ειδικέ αναπηρίες γιατί στα 87 εκατομμύρια καταλαβαίνετε ότι με την αύξηση του προσδοκίμου της ζωής έχουμε όλο και περισσότερο γυναίκες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε προκειμένου να στηρίξουμε τις γυναίκες αυτές με ειδικέ ανάγκες. Το δεύτερο σημείο το οποίο προτείνω στη γνωμοδότηση είναι η σημαντικότατη ανάγκη διάγνωσης αλλά και γρήγορων ε, λύσεων που θα επιτρέπουν στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρίες να είναι αυτόνομα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η ε, καθυστερημένη διάγνωση προκαλεί προβλήματα στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην ίδια την αυτονομία αυτών των ατόμων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η ανάγκη διάγνωσης, έγκαιρης διάγνωσης. Τρίτο σημείο. Λέω ότι πολύ συχνά είναι οι μητέρες αυτές οι οποίες λαμβάνουν τη φροντίδα των παιδιών με αναπηρίες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνέχεια στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε ένα πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας για αυτές τις γυναίκες, προκειμένου ο επιπλέον αυτός φόρτος εργασίας που προέρχεται από τη φροντίδα των αναπήρων παιδιών να ληφθεί υπόψη. Σήμερα το πρωί στη συζήτηση που είχαμε είπατε ότι θα πρέπει να συμφιλειωθεί η οικογενειακή και η επαγγελματική ζωή. Πολύ ωραία η πρόταση αυτή. Όταν όμως μιλάμε για παιδιά με αναπηρίες, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει στην γνωμοδότησή μας να υπογραμμίζουμε ιδιαίτερως αυτό το αίτημα. Επίσης, κάνω μία άλλη ρεαλιστική πρόταση που έχει να κάνει με τη ζωή των γυναικών αυτών που πρέπει να ασχοληθούν και να φροντίσουν παιδιά με αναπηρίες. Πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξουν την ιδέα αυτή. Και προτείνω οι σύλλογοι ε, γονέων με παιδιά ή ανηλίκων με αναπηρίες, που πολύ συχνά τελικά είναι άτομα τα οποία τα αντιλαμβάνουν οι γυναίκες, θα πρέπει λοιπόν να εμπλέκονται περισσότερο προκειμένου να γνωρίζεται περισσότερο η εμπειρία των γυναικών αυτών έτσι ώστε να υπάρχουν ε, λιγότερο αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική τους ε, σταδιοδρομία. Να υπάρχει λοιπόν μια επικύρωση της αποκτηθήσεως αυτής πείρας. Μιλάμε για επικύρωση διαφόρων δεξιοτήτων, διαφόρων επαγγελματικών προσόντων. Εγώ αυτό που ζητώ στο σημείο αυτό της γνωμοδότησης είναι οι γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν σε συλλόγους γονέων με παιδιά με αναπηρίες να χαίρουν μια επικύρωσης της αποκτηθήσης αυτής πείρας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν κάναν τη δουλειά αυτή οι γυναίκες αυτές, θα έπρεπε το έργο αυτό να τον αλάβουν τα κράτη οι εθνικές αρχές. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απόλυτα δίκαιο να αναγνωρίσουμε την αποκτηθή σε αυτή πείρα στην καριέρα τους. Στο σημείο 5 της γνωμοδότησής μου λέω ότι ε, είναι πολύ σημαντική η, ε, το ποσοστό των γυναικών με αναπηρίες στο γενικότερο φαινόμενο της γύρασης του πληθυσμού. Λέω ότι όλο και περισσότερο υπάρχουν ε, γυναίκες με αναπηρίες που γίνονται συχνά θύματα βίας. Η βία αυτή εκφράζεται όλο και περισσότερο κατά των γυναικών με αναπηρίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ως προς αυτό μια συγκεκριμένη πολιτική. Αναφέρουμε επίσης σε πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις γυναίκες με αναπηρίες να συνεχίσουν τις ε, σπουδές τους, ε, γιατί ε, πολύ συχνά οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδέ τους και κατά αυτόν τον τρόπο δεν καταφέρνουν στη συνέχεια να βρουν μια θέση εργασίας. Κάνω λοιπόν κάποιες πολύ συγκεκριμένε προτάσεις στη γνωμοδότηση αυτή προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες και προκειμένου να γνωριστεί η συμμετοχή των γυναικών όσον αφορά την φροντίδα ατόμων με αναπηρίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Προτού δώσω το λόγο στην κυρία Γκουρμάη, την πρώτη μας ομιλήτρια, σας πενθυμίζω για μια ακόμη φορά ότι θα πρέπει να είστε σύντομοι στις σας. Ευχαριστώ. So, uh, concerning... Uh, Τώρα, όταν μιλάμε για 80 εκατομμύρια ανάπηρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι φροντίζοντες είναι οι γυναίκες πολλές φορές χωρίς αμοιβή γιατί δεν είναι επαγγελματίες ούτε έχουν ασφάλιση κοινωνική η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να καλύψει αυτές τις γυναίκες ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την σύνταξη Η φτώχεια, η ανεργία είναι πολύ σημαντικά θέματα όταν μιλάμε για μόνες γυναίκες με ανάπηρα παιδιά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα της σχετικής έκθεσης εδώ. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και η ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται στην EU 2020. Να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να πετύχει η στρατηγική 2020 χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών και οι γυναίκες δεν μπορούν να ε, συμμετέχουν ως φροντίζοντες αν δεν αναγνωριστεί η δουλειά τους καλύτερα. Στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δύο φύλλα και να δίνουν αξιόπιστα στοιχεία για τους παρέχοντες φροντίδα. Δεν είναι πολλά αυτά. Η νοηματική γλώσσα τέλος πρέπει να αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας αναγνώρισης. Ευχαριστώ κυρία Γκουρμάη, κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος κυρία Σμάινερ που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Ε, θέτω τα εξή ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σαρτιέ καταρχήν και ως Επιτροπή Γυναικών, επειδή η Επιτροπή μας καταπολεμεί τις διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών και πολλά πολλές ανισότητες που αντιμετωπίζουν και μειονεκτήματα είναι σημαντικό να τονίσουμε τη θέση των αναπήρων γυναικών που δεν έχουν μόνο τα προβλήματα ως γυναίκες αλλά αντιμετωπίζουν και ως ανάπηροι διακρίσεις και γι' αυτό είναι διπλό το πρόβλημα. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τις ανάπηρες γυναίκες ε, έχει πολλά εμπόδια στην στρατηγική 2020 ε, έχουμε ποσοστό απασχόληση ως στόχο 70% αλλά δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε χωρίς πρόσβαση στην αγορά, διασφάλιση της πρόσβασης θα πρέπει να έχουν πραγματική ευκαιρία να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους. Πολλές φορές αυτό δημιουργεί απογοητεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προς συμφέρον μας να δουλέψουμε σκληρά για καλύτερη ενσωμάτωση των αναπήρων γυναικών και ανδρών που είναι το ένα έκτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Σημαντικό βήμα είναι να ενισχύσουμε την κινητικότητα των αναπήρων πολλοί αποκλείονται από την εκπαίδευση και από την εργασία γιατί έχουν μειωμένη κινητικότητα και δεν μπορούν να πάνε στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό χρειάζονται ειδικέ δράσεις και στρατηγικές για καλύτερη ενσωμάτωση των αναπήρων ανδρών και γυναικών που πολλές φορές είναι θύματα διακρίσεων που είναι αποτέλεσμα προκαταλήψεων και άγνοιας. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για τις ανάγκες και τα προβλήματα των αναπήρων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παρβάνοβα. Και εγώ είμαι σκιώδης και είμαι ομιλήτρια, θα είμαι πολύ σύντομη. Ελπίζω ότι μαζί με την εισηγήτρια και τη σκιώδης θα μπορέσουμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Σύντομα θέλω να πω το εξής. Εδώ μιλάμε για γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις σε δύο επίπεδα πρώτον λόγω του φίλου και δεύτερον ε, λόγω της αναπηρίας. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα δράσης Πιστεύω ότι το πρόγραμμα δράσης λοιπόν της Κομισιόν χρειάζεται περισσότερα μέτρα. Πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν για τους ανάπηρους άνδρες και γυναίκες. Θα πρέπει να μπορούν 100% να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, τίποτα λιγότερο. Πρόκειται για ανθρώπινο δικαίωμα ανθρώπων που έχουν αναπηρία. Βεβαίως πρέπει να έχουν και εκπαίδευση και δυνατότητα απασχόλησης να πηγαίνουν και σε, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αναψυχής όπως κάνουμε όλοι μας. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι πολύ συχνά σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε γυναίκες να αναλαμβάνουν την κυρία ευθύνη ανάπηρων παιδιών και μελών οικογενείας με αναπηρίες επίσης. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πιο προσεκτικά την κατάσταση στα κράτη-μέλη όπου έχουμε δει μια στροφή στην νοοτροπία όπου το κράτος έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να είναι οι γυναίκες μόνο υπεύθυνε γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχει κάποια προσωπική, κάποια βοήθεια, ένας βοηθός που εργάζεται και απασχολεί το πρόσωπο με αναπηρία. Και ο βοηθός είναι τα χέρια και τα πόδια του αναπήρου προσώπου και το βοηθεί να γίνει κινητικότερο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι ρόλοι σε κάποια κράτη-μέλη και πρέπει να πω ότι αυτή είναι η καλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα του κράτους ευημερία που έχουμε δει. Γιατί έτσι μπορούν οι ανάπηροι να συμμετέχουν σε μια φυσιολογική ζωή στην κοινωνία με τη βοήθεια αυτού του προσωπικού βοηθού. Υπάρχουν παιδιά που είναι σε αναπηρικά αμαξίδια και πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία μαζί με άλλα παιδιά με τη βοήθεια του βοηθού τους και συμμετέχουν και σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ζουν μια φυσιολογική ζωή. Γίνεται αυτό το πράγμα και θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει και να προσπαθήσει να ακολουθήσει τα παραδείγματα κάποιων κρατών μελών. Ξέρω ότι αυτό είναι ευθύνη κρατών, των κρατών μελών, όταν πρόκειται δηλαδή για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Αλλά χρήσιμο είναι να αναδειχθούν τα χρήσιμα παραδείγματα για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και τώρα η κυρία Πλάμ και μετά η κυρία Φιγκερέιδο. Ναι. Για ένα λεπτό να συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τις προτάσεις που κάνετε στην γνωμοδότησή σας. Διάβασα τον κατάλογο των δράσεων της Επιτροπής και θέλω να υπογραμμίσω ότι κάλλιστα μπορεί να συμπεριληφθεί η έμφυλη διάσταση σε όλες τις ε, δράσεις της στρατηγικής. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή και τα κρατη να εξετάσουν την έμφυλη διάσταση σε όλες τις επερχόμενες δράσεις. Κατόπιν, τονίζεται ότι οι γυναίκες με αναπηρίες υποεκπροσωπούνται στην δημοκρατική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων εν γέννη. Επίσης, οι γυναίκες που έχουν ψυχολογική αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους κατάχρησης από ότι οι άντρες με, τα, με τις αντίστοιχες αναπηρίες ή οι γυναίκες χωρίς αναπηρίες. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή, πρέπει να ζητήσουμε δηλαδή και τα κράτη-μέλη ακόμη περισσότερο, να αναγνωρίσουν το φύλλο ως μια σημαντική διάσταση για τα άτομα με αναπηρίες σε ό,τι αφορά τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Και ίσως και άλλα. Δεν ξέρω. δεν είδα στην ε, ιστοσελίδα της Επιτροπής αν η ανακοίνωση είναι και σε άλλα format. Audio, δηλαδή ακουστικά ή με το σύστημα Braille. Δηλαδή να μπορούν να γίνουν κατανοητά τα κείμενα αυτά από άτομα με αναπηρίες. Μπορεί και να μην είδα. Ίσως να μας τα πει ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Δεν το είδα. θα έπρεπε να είναι σε όλες τις μορφές format για οι πληροφορίες για να είναι διαθέσιμες. Μιλήσαμε για την προσβασιμότητα ως πρώτη βράση στη στρατηγική. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέντο, πρόεδρε. Ήδη η εισηγήτρια αναφέρθηκε σε πολλά σημαντικά θέματα και πολλές διαστάσεις. Θέλω να επαναλάβω ωστόσο κάτι που είπα προηγουμένως για τον προπολογισμό. Την ανάγκη να αυξήσουμε τη συγχρηματοδότηση για τις ενώσεις που δουλεύουν στον χώρο αυτό και που ζητούν χρηματοδότηση. Και στον τομέα αυτό δεν θα έπρεπε να τις επιβάλλουμε συμμετοχή χρηματοδότηση άνω του 10% του συνολικού προπολογισμού. Θα έπρεπε λοιπόν να προβλέψουμε από τώρα μία σχετική πρόταση. Ήθελα να την υποβάλω, αλλά ήθελα να σας το πω. Κάτι ακόμα. Το θέμα της απασχόλησης. Ήδη υπάρχει διάκριση των γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση. Όταν η γυναίκα είναι και ανάπηρη, η ανισότητα επιδεινώνεται. Το είπε και η συγκήτρια και είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Πρέπει να υπάρχουν θετικά μέτρα με κατάλληλη χρηματοδότηση. Η ίδια η Κομισιόν πρέπει να δώσει παράδειγμα. Με προτάσεις που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις και ρυθμίσεις για την καταπολέμηση αυτής της διπλής διάκρισης των ανάπηρων γυναικών στην πρόσβαση στην εργασία. Ε, Χρειάζεται λοιπόν και χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπο τη επιτροπή έχει το λόγο. Ή εκπρόσωπο τη επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση και για όλε αυτέ τι παρεμβάσει που ακούσαμε σήμερα που αναφέρθηκαν σε πολλά ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά και ευθυγραμμίζονται και καλύπτονται τελικά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική αναπηρίας για την επόμενη δεκαετία. Η στρατηγική αυτή έχει ως βάση την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τον Ιανουάριο δεσμεύεται ως προς τη σύμβαση αυτή και την έχει υπογράψει μαζί με τα κράτη-μέλη η διάσταση του φύλου αναγνωρίζεται σε αυτή τη σύμβαση και μάλιστα προβλέπεται στη σύμβαση αυτή και ένα επιπλέον μέσο προκειμένου στον, στη διάσταση αναπηρίας να έχουμε και τη διάσταση του φύλου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να σας πω ότι ε, όσον αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και όσον αφορά τα δεδομένα. Η στρατηγική για την αναπηρία συνδέεται πολύ με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και του στόχους που τίθενται εκεί, ιδίω όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας. Και σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει στο δείκτες και δεδομένα προκειμένου να έχουμε καλύτερη αναγνώριση των ατόμων και των γυναικών ιδιαίτερα με αναπηρίε, σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει για την απασχόληση, την παιδεία και την μείωση της φτώχειας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί το κενό αυτό γνώσης που υπάρχει στα κράτη-μέλη και το κενό δεδομένων, την απουσία δεδομένων και θέλουμε να υποστηρίξουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη σε αυτές τις προσπάθειες. Θα έχουμε λοιπόν τα δεδομένα τα οποία θα κατανέμονται με βάση το φύλλο όπου θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις αναπηριών, αναπηριών γυναικών και ανδρών και θα έχουμε και δεδομένα έπειτα για τον γενικό πληθυσμό, για τον ευρύ πληθυσμό. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της ε, ανακοίνωσης για την στρατηγική, αν είναι προσβάσιμη η ανακοίνωση αυτή και σε άλλους μορφότυπους, κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί και με εναλλακτική μορφή. Θα το διερευνήσω και θα έρθω σε επαφή μαζί σας για να σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος. Δίνουμε το λόγο στην συγκήτριά μας την κυρία Μωράν Σαχτιέ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, για τη συμβολή σας. Θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, προτείνοντας ως το δυνατόν πιο συμβαστικές τροπολογίες με τις οποίες θα μπορούσατε να συμφωνήσετε περισσότεροι. Βλέπω ότι ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις περιπτώσεις ε, διπλής ε, διάκρισης, γυναίκες δηλαδή με αναπηρίες και η Πρόεδρος και η κυρία Φιγκερέδο και η κυρία Παράνοβα και πολλοί άλλοι μίλησαν για το ζήτημα αυτό. Σημειώνω επίσης την βούλησή μας να ενσωματώσουμε περισσότερο τις θεραπείες μάλλον τις γυναίκες που έχουν αναλάβει τα άτομα με αναπηρίες. Η κυρία Σένσον Γκουρμά αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό και βλέπω ότι θέλετε περισσότερα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τα άτομα αναπηρίες αναφύλλω και να υπάρχει μια διασταύρωση αυτών των δύο δεδομένων. Αναφερθήκαμε επίσης και στα δημοσιονομικά προβλήματα και καταγράφω και την πρόταση της Ιλντα Φιγκερέιρο, την επανδιατύπωση της πρότασής της θα προσπαθήσω λοιπόν να λάβω υπόψη όλες αυτές τις ε, προτάσεις και με την δική σας σύμφωνη γνώμη θα σας προτείνω τροπολογίες που θα λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές και με τις οποίες ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 4 Μαΐου θα ψηφίσουμε στις 25, στις 16 Ιουνίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο στη μέση διάταξη. Ευγνωμοδότηση προς την Επιτροπή Απασχόλησης και αυτή η προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Τσέσκοβα είναι η συγγήτρια, τη δίνω μέσα στο λόγο και απευθύνω εκ νέου έκκληση να είστε συνθετικότατοι όλοι και όλες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας πω ότι ετοίμασα κάποιες σελίδες ε, για να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα την κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ένωση. Η συζήτηση για την έκθεση Κράτσα ήταν μεγάλη και ενδιαφέρουσα, οπότε θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνθετικά τα σχόλιά μου. Εμείς ετοιμάζουμε γνωμοδότηση, αλλά η αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Η ελεύθερη κυκλοφορία και η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μάλιστα συμβάλλει και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα γραφειοκρατικά και δυτικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Και η γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης ε, ασχολείται σημαντικά με το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, ε, δεν υπάρχουν έρευνες ειδικά για την κοινωνικότητα των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλειστικά δηλαδή. Από την έκθεση ωστόσο προκύπτουν πολλές δηλώσεις που αφορούν ακριβώς την έμφυλη διάσταση. Η κοινωνικότητα προφανώς εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, την προσωπική εμπειρία, την εκπαίδευση και οι διάφορε ε, μελέτες που είναι στη διαθέσή μα δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε επίπεδο κινητικότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες μετακινούνται συχνότερα, πολύ συχνότερα από τις γυναίκες, για επαγγελματικούς λόγους 44% των ανδρών ενώ 7% των 27% ε, των γυναικών μόνο. Και οι περισσότερες, τις περισσότερες περιπτώσεις αυτές είναι γυναίκες που συνοδεύουν τον σύντροφό του στη νέα θέση Το ποσοστό αυτό, το χαμηλότερο ποσοστό κινητικότητας των γυναικών οφείλεται εν μέρη και στην μικρότερη γενικότερη παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασία και εξαρτάται από τι ανισότητε ε, αμοιβή. Σύμφωνα με τι υφιστάμενε μελέτε, η κινητικότητα των γυναικών στηρίζεται σε μικρότερες προσδοκίες. Άρα ο στόχος δεν πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, ε, δηλαδή να πάει κάπου αλλού για καλύτερη δουλειά. Στις γυναίκες ε, παίζουν και, άλλες, ε, και άλλοι παράγοντες ρόλο. Φερρυπίν, ένταξη σε κοινωνικά δίκαια, δίκτυα, συγγνώμη, δυνατότητα σχολείων ή υποδομών για τα παιδιά Κάτι, ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες και οι άνδρες που μετακινούνται. Η ανεπαρκής ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που θα έχουν στη νέα χώρα. Πολύ συχνά δεν γνωρίζουν ποιες δυσκολίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν π.χ. γιατί αλλάζει το σύστημα κοινωνικής ε, προστασίας από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα και άρα περιορίζονται οι δυνατότητες ένταξης των εργαζομένων επειδή δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Κατόπιν. Υπάρχει η έκθεση της Επιτροπής για την υλοποίηση της Οδηγίας 38 του 2004 για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ένωση και το δικαίωμα και την ελευθερία κυκλοφορία. Στην ανακοίνωση αυτή για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν είναι ικανοποιητική η εφαρμογή της οδηγίας για τις γυναίκες και μάλιστα η έκθεση παρουσιάζει μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη που καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία Στη γνωμοδότησή μου εγώ τονίζω τρία βασικά θέματα που σχετίζονται με αυτά που ανέφερα προηγουμένω. Πρώτον, μιλάμε για την διαφορά αμοιβή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία. Ο παράγοντας αυτός πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις γνωμοδοτήσεις μας γιατί είναι ο κύριος λόγος που εμποδίζει την μετακίνηση των γυναικών για λόγους εργασίας. Δεύτερον, να κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη όταν ε, οι εργαζόμενοι μετακινούνται με σύζυγους, συντρόφους και παιδιά να παρέχονται κατάλληλες υπηρεσίες σε αυτούς. Και εδώ γίνεται, ο λόγος, γίνεται λόγος και για συντρόφους. Όχι μόνο για καταχωρημένες δηλαδή ενώσεις, αλλά για κάθε άτομο με το οποίο υπάρχει μία, ε, μία ε, σχέση μακροχρόνια ε, του εργαζομένου και του συντρόφου. Τρίτον, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να παράσχουν πλήρης πληροφορίες, πλήρη ενημέρωση στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους για να μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα στη νέα χώρα υποδοχής. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε. Προτού δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές, θα ήθελα να σας πω το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το διαθέσιμο χρόνο. Επομένως θα έχετε ως ανώτατο όριο τα δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Νότερα Λόβα. Θα μιλήσω αγγλικά για να πάω πιο γρήγορα. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένη η γνωμοδότηση αυτή. Συνεργάστηκα μαζί με την εισηγήτρια και έχουν συμπεριληφθεί πολλές από τις παρατηρήσεις μου. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν με το τελικό κείμενο. Θα ήθελα να πω εξ ονόματος τη ομάδα των σοσιαλιστών ότι το ζήτημα το οποίο μας απασχολούσε περισσότερο είναι το flexicurity, ασφάλεια με ευελιξία ιδίως ε, όσον αφορά τις ε, γυναίκες που δουλεύουν οπέρ, ε, την κινητικότητα των περιπτώσεων αυτών. Ξέρω ότι μιλάμε για γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κάποια σύμβαση, δεν προβλέπεται υγειονομική κάλυψη ασφάλεια και αυτό προκαλεί πρόβλημα βέβαια πολλές φορές. Όσον αφορά τώρα Στου στους εργαζομένους αυτούς που κινούνται πολύ για την εργασία τους. Είπαμε ότι οι περισσότεροι είναι άντρες, υπάρχουν όμως και πολλές γυναίκες που τους συνοδεύουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι γυναίκες λοιπόν αυτές να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο στην ε, κοινωνική ζωή της χώρας στην οποία πηγαίνουν, να καταφέρουν να βρουν μια δουλειά, να καταφέρουν να αυτοολοκληρωθούν Ξέρετε ότι τίθεται και το γλωσσικό ζήτημα πολλές φορές όταν πηγαίνει κανείς σε μια ξένη χώρα και όταν προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή σε μια άλλη χώρα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί δυνατότητα και στους στις συντρόφους να μάθουν την ε, γλώσσα της χώρας αυτής, να έχουν επίσης πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχω αυτή τη στιγμή το χρόνο για να τα καλύψω και προφανώ υποστηρίζω την γνωμοδότηση αυτή. Σα ευχαριστούμε κυρία Πλούμα. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Μίλησε η προαλήσασα πολύ γρήγορα πριν για τους διερμηνείς. Αυτό έθιξε εγώ απλώς. να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση αυτή. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να τονίσω ένα φαινόμενο το οποίο είναι απόρρια αυτή τη κινητικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εγκαταλείπονται. Παιδιά που έχουν γονείς οι οποίοι εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό το στο οποίο κατοικούν τα παιδιά. Έχει εγκριθεί ένα σχετικό ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένουμε τώρα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το ζήτημα. Πιστεύω πάντως ότι τουλάχιστον σε αυτή τη γνωμοδότηση θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα καταστρεπτικά για τις οικογένειες, ιδιαίτερα επιβλαβή για τα παιδιά εκείνα τα οποία αποχωρίζονται τους γονείς τους ή τα παιδιά εκείνα τα οποία πρέπει να ζήσουν πάρα πολύ μακριά από τους γονείς τους και να καλέσουμε μέσω της γνωμοδότησης αυτής τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση των παιδιών αυτών που τα έχουν αφήσει οι γονείς τους και να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν φυσιολογικά, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και ένταξη στην κοινωνική ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να γίνεται μια αναφορά στα παιδιά αυτά τα οποία θίγονται εξαιτία τη κινητικότητα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Δύο λεπτά σα πενθυμίζω ότι έχετε στη διάθεσή σα, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι το σχέδιο γνωμοδότησης είναι πολύ καλό. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση προκειμένου να εργαστούμε και εμεί περισσότερο. Μια σελίδα μόνο την οποία εμεί θα επεκτείνουμε πιστεύω έχετε θίξει κάποια πολύ κέρια σημεία, όπω για παράδειγμα ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι άντρε από ότι γυναίκε που χαίρουν του δικαιώματο κινητικότητα στα πλαίσια τη εργασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί εδώ πέρα ένα ισότιμο πεδίο συμμετοχής σε αυτού του είδους της αγοράς κινητικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβλέπονται όλα τα δικαιώματα άδεια μητρότητας για τις γυναίκες, καθώς επίσης και το να υπάρχει υπηρεσία φροντίδας για τα παιδιά, να υφίσταται και το δικαίωμα άδειε πατρότητας προκειμένου οι οικογένειες με παιδιά να μπορούν να χαίρουν του δικαιώματος αυτού κινητικότητας. Η κυρία Πλάμα αναφέρθηκε στα παιδιά αυτά τα οποία αποχωρίζουν τους γονείς τους. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε στη γνωμοδότηση. Ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για το πρόβλημα αυτό και η λύση θα ήταν ενδεχομένως να μπορέσουν οι οικογένειες με παιδιά να ασκήσουν πολύ πιο εύκολα τα δικαιώματά τους. Οι γυναίκες βρίσκονται σε πολύ πιο ευάλωτη θέση το ότι πολλές φορές ε, δεν καταφέρνουν οι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν σε κάποια άλλη χώρα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Οπότε πολλές φορές δεν καταφέρνουν να υποφεληθούν των δικαιωμάτων τους σε άλλες χώρες και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. Οι σύντροφοι τώρα, οι σύζυγοι. Καταρχάς, έχουμε και τους συντρόφους αυτούς στα πλαίσια μιας ομοφιλοφιλικής σχέσης και αυτοί δεν καταφέρνουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και θα πρέπει να γίνεται μια αναφορά και στους διεμφιλικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Σε τρία σημεία αναφέρονται πολλά πράγματα γιατί αναφέρονται τα περισσότερα προβλήματα των αναπηριών. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούσαμε, συμφωνώ βέβαια με όλους όσους μίλησαν ήδη, αλλά δεν θα μιλήσω μόνο για τα παιδιά, αλλά και τις γυναίκες, τις γυναίκες που εγκαταλείπονται γιατί συνήθως είναι οι άνδρες κινητικοί, αλλά λείπουν για μήνες από το σπίτι. Και συχνά οι γυναίκες είναι άνεργες, γιατί περνάμε οικονομική κρίση, αλλά δεν μπορούν να τους ακολουθήσουν και δεν έχουν πληροφορίες για ε, τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχουν. Οπότε είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην ανάγκη να ενημερωθεί ο κόσμος. Σήμερα με την υψηλή τεχνολογία που υπάρχει στον κόσμο εύκολο είναι να φτιάξουμε ένα φυλάδιο για τα βασικά δικαιώματα ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και να πάνε σε έναν άλλο τόπο. Αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας. Σήμερα για να βρει κανείς τη σωστή πληροφορία πρέπει να επισκεφτεί 10 διαφορετικούς δικτυακούς τόπους και δεν θα καταλάβουν ίσως όλοι. Υπάρχει και ο γλωσσικός φραγμός και τα παιδιά και οι γυναίκες πλήττονται. Τώρα για τους μισθούς. Δεν ξέρω αν σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά στα μισά τουλάχιστον οι μισθοί θεωρούνται εμπιστευτικοί απέναντι σε τρίτους. Και στην Εστονία αυτό ισχύει και για το δημόσιο τομέα. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα αν δεν ξέρουμε τι κερδίζουν οι συναδελφοί μας. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να είναι εμπιστευτικά τα στοιχεία αυτά, αλλά να υπάρχει πρόσβαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Οβίρ. Η κυρία Τσέσκοβα, δύο λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τα εντάξω όλα αυτά στην έκθεση, στη γνωμοδότηση αλλά επειδή θεωρητικά συμφωνούμε όλοι. Με εκπλήξατε λίγο με τα παιδιά που εγκαταλείπονται, που μένουν πίσω. Έχω δύο παιδιά και δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα πήγαιναν οι γονείς στη δουλειά αφήνοντα πίσω τα παιδιά. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο για μένα. Στις αναλύσεις μου του θέματος ε, μίλησα και με συμβούλους από το δίκτυο EUREST που αφορά και θέσεις που προσφέρονται στο έδαφος της Ένωσης. Και υπάρχει πληροφόρηση σχετική, υπάρχει ένα εγχειρίδιο με όλες τις πληροφορίες. Οπότε αναφέρονται και οι απαιτήσει και οι τα επιδόματα που μπορούν να δοθούν οι παροχές όταν μετακινούνται οι οικογένειες. Κρίμα που είχαμε τόσο λίγο χρόνο γιατί είχα ετοιμάσει και μια γνωμοδότηση με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που αποφάνθηκαν με πολύ σημαντικό τρόπο γιατί το δικαστήριο προχώρησε σε ορισμούς τι είναι ένα σύντροφος, τι, τα παιδιά κλπ. Ελπίζω ότι αργότερα ή την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τσέσκοβα. Και εγώ ελπίζω να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για μια συζήτηση πάνω σε, αυτές τις, ε, σε αυτά τα θέματα. 3 Μαΐου, 25 Μαΐου στην Επιτροπή, 16 ε, Ιουλίου στην ε, Επιτροπή, τον Ιούλιο θα πάει στην Ολομέλεια. Κρίμα που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο σήμερα το πρωί, αλλά πρέπει να σπεύσουμε να πιάσουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, σημείο 11, το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δίνω το λόγο χωρίς άλλα, άλλο στην κυρία Κώστανη, συντάκτρια. Θα είμαι συνθετική. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση η έκθεση της ΛΥΜΠΕ γιατί είναι η πρώτη πραγματικά έκθεση με πρωτοβουλία της Επιτροπής με σαφείς ε, θέσεις για ζητήματα που αφορούν εν γέννη το οργανωμένο έγκλημα από διάφορες οπτικές γωνίες. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώ να υπάρχει μέσα στην έκθεση αυτή και η διάσταση του φύλου για πολλούς λόγους που γνωρίζουμε. μια ενημέρωση πρακτικού χαρακτήρα. Χτες έγινε συνάντηση των σκιωδών. Η συγγήτρια, κυρία Αλφάνο, άτυπα παρουσίασε 60 τροπολογίες για την έκθεσή της. Όλοι χρησιμοποίησαν χρόνο και η προθεσμία είναι η εξής αναβλήθηκε η ψηφοφορία στην Λίμπε και θα πάει στην Ολομέλεια, θα πάει στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Η Λίμπε έχει προθεσμία 20 Μαΐου, θα ψηφιστεί 19 Σεπτεμβρίου. Για μας πάμε για 4 Μαΐου τροπολογίες και 25 πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Αυτά σας το λέω γιατί έγιναν οι αλλαγές. Στην έκθεσή μου προσπάθησα να έχω 1400, 1400 χαρακτήρες. Έκοβα, έκοβα, έκοβα. Έκοψα λοιπόν τα βασικά θέματα που κατόπιν θα χρειαστεί να ξαναδιευρυθούν. Και σας λέω και τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις για τροπολογίες. Να τονίσω ωστόσο ότι επειδή η έκθεση της ΛΥΜΠΕ είναι εξαιρετικά εκτεταμένη, θα πρότεινα οι, οι τροπολογίε μα και το προτείνω στου συναδέλφου να περιοριστούν στις πολύ σημαντικέ για να μην βγουν πολλές τροπολογίε και μα τι πετάξουν έξω επειδή είναι πολλέ. Πρώτη παρατήρηση. Οι νέε γυναίκες είναι ένα μεγάλο τμήμα των θυμάτων του οργανωμένου εγκλήματος. Ιδίω σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά του προσώπου. Υπογραμμίζουμε λοιπόν ότι η πρώτη πρόληψη της εγκληματικότητας είναι κοινωνική ένταξη, μάχη κατά των ανισοτήτων. Τρίτο, οι γυναίκες είναι γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη είναι μειονότητα μεταξύ των εγκληματιών αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάποιες διαστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Φερρυπίν, την εκμετάλλευση θυμάτων εμπορίας ή ε, εμπόριων ναρκωτικών ή στις μαφιόζικες οργανώσεις όπου είναι και θύματα και ε, συνένοχοι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία μεγαλύτερη έμφαση στην διάσταση του φύλου, να υπάρξουν στοχοθετημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καμπάνια ευαισθητοποίησης μαζί με ΜΚΟ, βοήθεια στα θύματα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών ζητούμε την εφαρμογή της οδηγίας ε, κατά του, της εμπορίας, ιδίως το ρόλο του συντονιστή κατά του τράφικινγκ, γιατί να, δίνοντας, να δίνει δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου, ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία όλων των θυμάτων. Μην ξεχνάτε ότι κατά τη συζήτηση για το ΟΠΕ, είχαμε πει ότι η προστασία αυτή θα έπρεπε να επεκταθεί σε άλλο επίπεδο και στα θύματα, στους μάρτυρες και τα μέλη της οικογένειας θυμάτων οργανωμένου εγκλήματος πέραν της εμπορίας. Μια συγκεκριμένη παρατήρηση και ερώτηση μάλλον. Να σκεφτούμε ειδικού τρόπους προστασίας της ασφάλειας και οικονομικής ασφάλειας των γυναικών. Αυτό συμβαίνει σε πολλές ε, οργανώσεις, σε πολλές συμμορίες που θέλουν να εγκαταλείψουν το έγκλημα αλλά μπορεί να είναι εκτεθειμένες σε αντίπεινα. Επίσης, κυρώσεις για τους χρήστες υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, εμπορίας και ή εμπορίας ανθρώπων και τέλει την ε, ανάδειξη του ρόλου των γυναικών σαν ενεργού μαχητή της εγκλημα, κατά της εγκληματικότητας, δικαστίνες, ε, εκπαιδευτικοί, Κάποιες τροπολογίες τώρα που θέλω να υποβάλω είναι πρώτον το θέμα του Eurojust και της Europol να μην ξεχνάτε ότι στην Europol υπάρχει μια ετήσια έκθεση που πρέπει να περιλαμβάνει μια διάσταση των γυναικών. Να προωθήσουμε το ρόλο των γυναικών ε, και των ε, ενώσεων των οικογενείων των θυμάτων και να σκεφτούμε και ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για τις ενώσεις αυτές που έχουν συγκεκριμένα ζητήματα και όπου συχνά οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο. Το θέμα της ειδική προστασίας για το κυβερνοέγκλημα που εμπλέκει γυναίκες και ανηλίκους και τη δυνατότητα μορφών αποζημίωσης ιδίως για τους ανηλίκους λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνικό χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα δίκημα μπορεί να γίνει σε μια χώρα, η ζημιά μπορεί να η βλάβη ο ομιλήτρια. Η βλάβη μπορεί να είναι σε μία χώρα, αλλά η αποζημίωση σε άλλη. Και κατόπιν το ρόλο των μορφών αποζημίωσης, όπως έλεγα προηγουμένως, όλων των γυναικών που καταγγέλουν και μπορούν να είναι εκτεθειμένες με τη σειρά του σε κάποια μορφή αντιπίνων. Βεβαίω περιμένω όλες τις προτάσεις σας. Πρόκειται για, μόνο μια, για μια μόνο πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Πρωτού δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα στην Επιτροπή μας, μια ομάδα φοιτητών από την Σουηδία που σπουδάζουν gender politics, πολιτικές όσον αφορά το φύλλο, από το Πανεπιστήμιο του Λούντ. Το λόγο αναφέρομαι στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Κώστα και μπορούμε να στηρίξουμε και το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Αλφάνο. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία σημεία στα οποία αναφέρθηκε η συγγήτρια. Όσον αφορά την πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος και εν γέννη του εγκλήματος, προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα και του σχεδίου δράσης της Στοκόλμης και της ανακοίνωσης για την εσωτερική ασφάλεια. Και, όπως και στο παρελθόν, ήδη έχουμε αναπτύξει πολλές δράσεις για την πρόληψη του εγκλήματος εν γέννη, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που άπτονται ιδιαίτερα της διάστασης του φύλου και συμφωνούμε με τις τρεις προτεραιότητες που βλέπουμε εδώ πέρα στην γνωμοδότηση. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο πρόγραμμα ISAC το οποίο προβλέπει χρηματοδοτική υποστήριξη ανά έργο, ανά σχέδιο προκειμένου να προωθηθούν πρωτοβουλίες κατά του οργανωμένου εγκλήματος και στην, στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων μπορείτε να δείτε τα σχέδια αυτά τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν. Θα ήθελα να αφαιρθώ επίσης και στην υποστήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, της το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την πρόληψη του εγκλήματος με την πρόθεση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. 750.000 ευρώ δώσαμε πέρυσι στο δίκτυο αυτό. Όπως γνωρίζετε, σε διάφορες νομικές προτάσεις που έχουμε κάνει, συστηματικά συμπεριλαμβάνουμε διατάξεις που έχουν να κάνουν με την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου εγκλήματος. Η συγγήτρια άλλωστε αναφέρεται στην οδηγία για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων. Και ως προς αυτό υπάρχει μία σημαντικότατη διάταξη για την πρόληψη του εγκλήματος αυτού. Επίσης, ε, στηρίζουμε την ε, ανάγκη ε, καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Συντοποιούμε ότι είναι κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα θύματα αυτού του εγκλήματος και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την έγκριση και δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της νέας αυτής οδηγίας με νέες ε, ρήτρε για την υποστήριξη των θυμάτων αυτών και για την πρόληψη του φαινομένου πορεία ανθρώπων. Τέλος, να αναφερθώ στην ανάγκη προστασίας των θυμάτων. Για το ζήτημα αυτό συμφωνούμε πλήρως όσα λέγονται εδώ στη γνωμοδότηση στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνταχθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου μία νέα ανακοίνωση δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή οι μάρτυρες και οι συγγενείς τους, καθώς επίσης και τα άτομα που συνεργάζονται με την αστυνομία. Θα φροντίσουμε όμως να προβλέψουμε μια προστασία για τα θύματα και τους μάρτυρες στο μέλλον. Και το, σε σχέση με την οδηγία του 2004 θέλουμε να επιλύσουμε και το ζήτημα αυτό το οποίο εκκρεμεί όσον αφορά την αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος. Ευχαριστώ. Eh, Κώστα, Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για τα θέματα αυτά που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Αυτό μπορεί να το ενισχύσουμε εδώ. Τα προγράμματα κατά του εγκλήματος. Είναι πολύ ωραίο που η αρμόδια γενική διεύθυνση εξετάζει το θέμα της προστασίας των μαρτύρων. Ελπίζουμε ότι όλα τα θύματα άμεσα και έμεσα του οργανωμένου εγκλήματος, όχι μόνο οι γυναίκες και οι ανήλικοι, αλλά και οι άλλοι, θα ωφεληθούν και ότι αυτό θα είναι μια έκθεση πλαίσιο. Χάρηκα λοιπόν που άκουσα την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ τη συντάκτρια. Όπως είπε και η ίδια, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για κατάθεση τροπολογιών από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. 4 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης, αντί για τις 20 Απριλίου, 25 Μαΐου ψήφος στην Επιτροπή, ψήφος ψηφοφορία στη Λίμπε 19 Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο θα πάει στην Ολομέλεια. Οπότε τώρα προχωρούμε στο επόμενο σημείο είναι το σημείο 12. Μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΑΦΕΤ και αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκού Εκδημοκρατισμού. Η αρμόδια συντάκτρια στην Επιτροπή μας είναι η κυρία Παπαδοπούλου, στην οποία δίνω αμέσω το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Παπαδοπούλου. Α, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη λόγω χρονικών περιορισμών. Χαιρετίζω την παρουσία της κυρίας Βερονίκ Ντεκάιζερ που είναι η συγγήτρια για το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ΑΦΕΤ για το θέμα αυτό της εξωτερικές πολιτικές για τον εκδημοκρατισμό. Ως η συγγήτρια από την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των Φύλων θέλουμε η Επιτροπή ΑΦΕΤ να ενσωματώσει κάποιες προτάσεις μας στο, στην πρόταση ψηφίσματος. Στο έγγραφο εργασίας της κυρίας Ντεκάιζερ υπάρχει ειδική μνήα των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να επικεντρώνουν στην ανάγκη εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες. Η γνώμη μου λοιπόν είναι πολύ σχετική σχετικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών υπέρ του εκδημοκρατισμού. Επίσης τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τις, τα κινήματα βάσης και την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτή είναι η ιδέα αυτό θέλουμε να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών για να έχουν παρουσία στις σοβαρές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το μέρος του κόσμου και όχι μόνο. Αυτό που θέλουμε να προβληθεί από τη δική μας την Επιτροπή Γυναικών είναι ότι θέλουμε μια συνολική στρατηγική της Ένωσης που θα θέτει προτεραιότητες συγκεκριμένες, είναι μακροπρόθεσμη προσέγγιση που θα διασφαλίσει την ισότητα των φύλων ώστε να μπει στην καρδιά όλων των κοινωτικών πολιτικών, προγραμμάτων, έργων, δραστηριοτήτων, ό,τι προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα ε, όταν μιλάμε για σχέσεις ε, μεταξύ Ένωσης και των χωρών. Σταθερότητα, συνοχή, ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά. Θέλουμε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το σημαντικό της ρόλο για να εξυγχρονίσει και να ενισχύσει θέματα ισότητας σε θεματικές προτεραιότητες και μέσα από τη χρήση συμμετοχικών προσεγγίσεων στο σχέδιο και ανάπτυξη των έργων, να δώσει έμφαση στην καταπολέμηση των στερεοτύπων κατά του φύλου και ε, να καταργήσει τη βία των γυναικών, τη διακρίσεις, εντάσσοντας τις γυναίκες ε, στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, επιτρέποντάς τις να είναι ενεργοί πολίτες. Πιστεύουμε ότι το 52% είναι οι γυναίκες που σύμφωνα με στατιστικές αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών. Οπότε ο ρόλος των γυναικών στη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων είναι σημαντικός. Η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα θα βοηθήσει πραγματικά και θα έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ειδικού προγράμματος των γυναικών. Τέλος, θέλουμε σε αυτό τα προγράμματα ισότητας φύλων να υπάρχει συστηματική πρόσβαση και αξιολόγηση, να διασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση, γιατί ακόμα και αν υπάρχει πολιτική βούληση υπέρ του εξυγχρονισμού, εκδημοκρατισμού, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Τέλος, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης προσπαθεί να προσλάβει περισσότερους άνδρες και γυναίκες και να έχει κατανομή 50-50 μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο επικεφαλής αντιπροσωπιών. Ελπίζομαι ο στόχος να επιτευχθεί γιατί αν δεν δούμε γυναίκες σε θέσεις με επιρροή όπου λαμβάνονται αποφάσεις δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αλλαγές. Αυτές είναι οι συστάσεις μας λοιπόν. Είμαι θα ευτυχής που είναι εδώ η κυρία Ντεκάιζερ. Ελπίζω να ενσωματωθούν αυτά στην έκθεση της Επιτροπής σας αφέτε. Δυστυχώς οι τροπολογίες θα έπρεπε να κατατεθούν σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα που έλεγε η προθεσμία. Είναι λίγο ηρωνικό να συζητάμε το θέμα, να ακούμε τις ιδέες και να, ε, ε, να έχει λήξει ο χρόνος προθεσμία κατάθεσης. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί χρόνος, να υπάρξει μια αναβολή, να μας δοθούν δύο ώρες ακόμα, ώστε να ακούσουν σήμερα, να καταθέσουν, ας πούμε τρεις η ώρα το απόγευμα της ε, τροπολογίες. Αν γίνεται, αυτή την πρόταση ήθελα να σας υποβάλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζαμπόρσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω και εγώ με την ε, συντάκτριά μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους τροπολογίες, καλό θα ήταν να έχουμε προθεσμία στις 3 το απόγευμα. Κάποια γενικά σχόλια καταρχήν. Χαίρομαι που είναι και παρούσα η κυρία Ντεκάιζερ η έκθεση αποδεικνύει ότι υπάρχουν πολλές εμπειρίες στον τομέα του αναπτυξιακής δουλειάς. Ε, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή α, καλύπτει τις απόψεις και τα αισθήματα πολλών ευρωβουλευτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, αναλάβει ενεργό δράση εις ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες. Οι βουλευτές σε πολλές εκθέσεις, για παράδειγμα σε σχέση με την Βόρεια Αφρική, τη Λευκορωσία, ε, κατέστησαν, ε, ε την προσοχή στους εκπροσώπους της Κομισιόν ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες και να προβλέπονται και ανάλογες κυρώσεις. Η έκθεση αυτή θεωρώ ότι είναι μια κατεπίγουσα έκθεση του Κοινοβουλίου. Ο στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα βήματα. Τώρα, για τη γνωμοδότηση της δικής μας της Επιτροπής. Ευχαριστώ την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης διότι αναφέρει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στους άνδρες και στους γυναίκες διαφυλάσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα σημεία 1 και 2 η συγγήτρια μιλάει για την πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομίζω ότι πρόκειται για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε τρίτες χώρες. Ίσως θα ήταν καλό να, βάλω, να, να, να μην μιλήσουμε για επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για τρίτες χώρες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην ε, διαφύλαξη και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τρίτο κόσμο. Θα ήταν καλύτερο να μην μιλήσουμε με ιδεολογικούς όρους. Καλύτερα θα ήταν να μιλήσουμε για την ισότητα των φίλων. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν προβλήματα ενδεχομένως με τη διατύπωση. Πρέπει να είναι προσεκτική όμως η διατύπωσή μας και να μην ακούγεται τυποποιημένη. Είναι ασυνέπεια το ότι σε πολλές χώρες, στο Κονγκό για παράδειγμα, στη δημοκρατία του Κονγκό παραβιάζονται ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμείς δεχόμαστε το χαρακτηρισμό αυτών των χωρών. Ε, νομίζω ότι είναι καλό λοιπόν και αυτό που προτείνετε κυρία Πρόεδρε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπε η συντάκτριά μας σε σχέση με την ε, στενή προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών πραγματικά μας λυπεί ότι είναι τόσο πιεστικά τα περιθώρια, αλλά μας ενδιαφέρει σε σχέση με τις προθεσμίες που έθεσαν στην ΑΦΕΤ. Αυτό το είχαν βάλει από παλιότερα στην ημερήσια διάταξη και έπρεπε να γίνει αλλαγή για άλλους λόγους. Κατ' εξαίρεση, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα, ώστε να κατατεθούν τροπολογίες μέχρι τις 2 σήμερα κατ' εξαίρεση θα έχετε αυτή την ευκαιρία. Αλλά δύο το απόγευμα ε, χωρίς άλλη αλλαγή. Κυρία Πλάμ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ για τη γνωμοδότησή της, ε, τη συναδελφό κυρία Παπαδοπούλου και να ευχαριστήσω την κυρία Ντεκάιζερ για την παρουσία της εδώ. Είχε μια μακρά εμπειρία στο θέμα αυτό των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Πιστεύω ότι όντως πρέπει να ενισχύσουμε την διάσταση του φίλου. Θυμηθείτε τι έγινε σε αραβικές χώρες, την Τινησία και την Αίγυπτο ιδίως πρόσφατα. Οι γυναίκες είχαν βγει στο δρόμο και αγωνίζονταν για τα δικαιώματά τους. τώρα αγωνίζονται για την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. και για την αύξηση των δικαιωμάτων ε, της ισότητας. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ξανά και περισσότερο ότι χρειαζόμαστε την πλήρη συμμετοχή της γυναίκας σε όλους τους τομείς την ασφάλεια και την ειρήνη για την ενίσχυση της ε, Πρόληψη των συγκρούσεων και τη διασφάλιση βιώσιμης ειρήνη. Να πω επίσης ότι όχι μόνο στον τομέα αυτό αλλά και στο διεθνές εμπόριο πρέπει να περάσουμε το mainstreaming στο φύλλο, του φύλλου διότι χρειαζόμαστε παρουσία των γυναικών σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις. Να τονίσω επίσης την ανάγκη προοπτικής του φύλου στην εφαρμογή των καθηγητών γραμμών για τις οχοθετημένες θέσεις υπέρ των δικαιωμάτων των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων όπως τα δικαιώματα των παιδιών, την της ε, των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστώ. Τελειώσανε. Κύριε Παπαδοπούλου για τα τελικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λέω ότι χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω την υπεύθυνη εισηγήτρια της Επιτροπής ΑΦΕ, την κύριο Ντικέιζερ. Θέλετε και το λόγο. Ε, το θέλω, πρόεδρε. Γιατί ήρθα για να σας ακούσω. Αλλά να πω κι εγώ δύο λόγια. Κύριος, πόσο υπάρχει ένα θετικό απρόοδο για τις εργασίες σας στην έκθεσή μου. Ε, μία φορά μόνο αναφέρθηκα στο θέμα των γυναικών γιατί ξέρω ότι ετοίμαζε γνωμοδότηση Επιτροπή Γυναικών και άρα έπρεπε να υιοθετήσω ό,τι περισσότερο μπορούσα από τη γνωμοδότηση αυτή. Για την ανάγκη δηλαδή να θέσουμε την ισότητα, το φύλλο στο κέντρο της πολιτικής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της εξωτερικής πολιτικής με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη. Αυτά μόνο. Σταματώ εδώ. Πρόκειται για να σημαντικό, για μια σημαντικό ορόσημο. Είπαμε ότι οι γυναίκες, το ακούστηκε αυτό, οι γυναίκες αγωνίζονται για να μετάσχουν στο δημοκρατικό κίνημα. Ε, εν γέννη, μετά αποκλείονται από τη διαδικασία αυτή. Αγνοούνται στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι χώρες με τις οποίες έχουμε πολλές σχέσεις και που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για την ελευθερία και τη δημοκρατία τους θα πρέπει να μην ξαναχάσουν τις γυναίκες τους. Ιστορική στιγμή λοιπόν. Θα υποδεχθώ με ανοιχτές αγκάλες τις προτάσεις της Επιτροπής σας. Δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτά που θα πείτε εσείς. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό η κυρία Γκουρμάη. Μα πρόκειται για ιστορική στιγμή, όπως είπε η φίλη μου η Βερονίκ, γιατί είχαμε και τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία ανασυγκρότησης εκεί και οι γυναίκες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία αυτή. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο υπήρχε τότε μια task force για τις γυναίκες για τη διάσταση του φίλου ήταν ακριβώς για το λόγο αυτό. Σε ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαδοπούλου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε μια νέα προθεσμία μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δέχομαι γραπτός λοιπόν τις παρατηρήσεις σας φαίνεται τελικά ότι η ισότητα των φύλων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ζήτημα προτεραιότητας, ιδίω στις τρίτες χώρες, τη στιγμή αυτή που βλέπουμε ότι υπάρχει τόση μεγάλη κοινωνική αναστάτωση και υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διεκδικούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι γυναίκες έχουν και αυτές το δικαίωμα να συμμετέχουν στο μηχανισμό λήψη αποφάσεων, να συμβάλλουν ενεργά στο μέλλον των χωρών τους, και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι η κυρία Ντεκάιζερ θα συμπεριλάβει τις προτάσεις αυτές της γνωμοδότησης στη δική της την έκθεση. Διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση Τη κύρια Ντεκάιζερ και αναφερόμενη η κυρία Ντεκάιζερ στου βασικού πυλώνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον μου κάνει εντύπωση αυτό που είπα ότι δεν, θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε σφάλματα κρίση στο μέλλον. Και κάθε φορά που υπάρχουν παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε πρόκειται από τη μία ή την άλλη χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση θα πρέπει να έχει ε, διακριτική μεταχείριση, δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβάλλει κυρώσεις, να αγωνίζεται για τις ε, ευρωπαϊκές ε, παγκόσμιες αρχές και να τις προωθεί και να επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Η διάσταση λοιπόν του φύλου θα πρέπει να υπάρχει και στην τελική έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό ζητάμε μέσω της γνωμοδότησής μας. Σας ευχαριστώ. E- Προθεσμία για τις τροπολογίες έλεξε όπως είπαμε Οι τροπολογίες που θα σταλούν πριν τις 2 το μεσημέρι σήμερα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία. Ευχαριστώ όλες σας και όλους σας για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρωινή συζήτηση. Εξίσου ενδιαφέρουσα θα είναι η απογευματινή συνάντησή μας, όπου έχουμε μία ακρόαση που ξεκινά στις 3 να είστε όλες εδώ. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ και τους διερμηνείς.